Äh, Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε με τις συνεδρίες της Επιτροπής και την ακρόαση της εκτελεστικής διευθύντριας της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ΕΦΣΑ, στην Πάρμα. Η κυρία Κατρίν Ζεσλά Λανέλ ε, είναι μαζί μας και την καλωσορίζουμε. Δεν είναι πρώτη φορά που έρχεται εδώ, αλλά σήμερα έρχεται για μια ιδιαίτερη περίσταση. Ήσασταν υπεύθυνοι της αίθουσα στην Πάρμα τα τελευταία πέντε χρόνια και την 1η Ιουλίου του 2011 λίγη η θητεία σας. Σύμφωνα με τον κανονισμό 178 του 2002 προβλέπεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση ένα κατάλογο υποψηφίων που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά από ανοιχτό διαγωνισμό θα υποβάλει μία πρόταση και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσει με την πρόταση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 7 Νοεμβρίου αποφάσισε να ανανεώσει τη θητεία της κυρίας Κατρίν Τζεσλα Λανεέλ για άλλα πέντε χρόνια και ο Επίτροπος Ντάλι έστειλε στην Επιτροπή μας μια αντίστοιχη επιστολή στις 25 Νοεμβρίου. Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στη σημερινή ακρόαση. Πρέπει να κάνουμε την ακρόαση και στη συνέχεια να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αυτό το οποίο θα στείλουμε ως επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συζητηθεί στη συνάντηση των συντονιστών μετά τη σημερινή ακρόαση. Όλοι γνωρίζουμε τη διαδικασία, αγαπητοί συνάδελφοι, από τις ακροάσεις των Επιτρόπων. Και σήμερα το πρωί αντίστοιχη ακρόαση θα γίνει φροντίζουμε και το χρόνο. Εγώ θα φροντίσω να τηρήσουμε τους κανόνες όσον αφορά το χρόνο. Ξεκινάμε λοιπόν με μια παρουσίαση της κυρίας Ζεσλά Λανέλ επί 10 λεπτά. Ποια είναι τα βασικά σημεία του προγραμματό σα, ποιε είναι οι προθέσει σα και το πρόγραμμά σα για τα επόμενα πέντε χρόνια. Στη συνέχεια θα λάβουν το λόγο οι συντονιστέ και θα ακολουθήσουν δύο γύροι συζητήσεων με τα υπόλοιπα μέλη τη Επιτροπής και στο τέλο άλλα πέντε λεπτά για την κυρία Ζεσλα Λενεέλ. Και έχουμε και το παιχνίδι πινκ-πονγκ των ερωτήσεων και απαντήσεων ένα λεπτό για μετά συμπληρωματικών ερωτήσεων και απαντήσεων. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως. Κυρία Ζεστιλά Νενέλ έχει το λόγο για την παρουσίαση του προγράμματός της για τα επόμενα πέντε χρόνια στην ΕΦΣΑ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, Είμαι πάντα ευγνώμων που μου δίνετε την ευκαιρία να έρχομαι εδώ και να μιλάω μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ανταλλάσσω απόψεις μαζί σας όσον αφορά τις δραστηριότητε της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων, την ΕΦΣΑ. Παρόλο που τα ευρετικά κείμενα αναφέρουν ότι έχουμε μια καθαρά επιστημονική αποστολή. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν ε, γενικότερα θέματα που απασχολούν την κοινωνία όσον αφορά την τροφική αλυσίδα και πρέπει και αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας στο έργο μας, όπως την ε, διαχείριση κινδύνου. Αυτή η αιτήσια ανταλλαγή απόψεων που έχουμε με το Κοινοβούλιο είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί μπορούμε να συζητάμε έτσι τις ε, εξελίξεις στην ΕΦΣΑ. Η δικιά σας στήριξη ήταν ε, πάντα πολύ σημαντική και μας βοήθησε να προχωρήσουμε στο τόσο σημαντικό έργο της ΕΦΣΑ που είναι η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών. Έχετε δείξει και τον Ιούνιο που μας πέρασε πόσο σημαντικό θεωρείται το έργο της ε, ΕΦΣΑ με την αντιπροσωπεία σας που ήρθε με την προεδρία του Τζο Λέινεν στην Πάρμα, στα γραφεία μας. Η επίσκεψή σας εκεί ήταν πολύ ενθαρρυντική για όλο το προσωπικό της ε, ΕΦΣΑ που συνεισφέρει στις δραστηριότητε τη ΕΦΣΑ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σα ευχαριστώ πολύ επίση και για τη στήριξή σα στην ΕΦΣΑ στον προπολογισμό του 2011. Το 2010 ε, αναθέσαμε δύο ανεξάρτητες μελέτες προκειμένου να μετρήσουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τις επιδόσεις της ε, ΕΦΣΑ τα τελευταία 8 χρόνια. Η πρώτη τέτοια έρευνα έχει να κάνει με το ευρωβαρόμετρο όσον αφορά το πώς αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές τον ε, κίνδυνο που έχει να κάνει με τα τρόφιμα. Και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες συνδέουν το φαγητό με τη γεύση και την απόλαυση και νιώθουν ότι προστατεύονται από το σύστημα ασφάλειας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σε σχέση με το από πού αντλούν τις πληροφορίες τους ε, οι καταναλωτές, διαπιστώνουμε ότι οι επιστήμονες έρχονται στην τέταρτη σειρά. Πρώτα έρχονται οι επαγγελματίες της υγείας, μετά η οικογένεια, μετά οι οργανώσεις καταναλωτών και τέταρτη οι επιστήμονες. Και τα δύο τρίτα θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό να εμπιστεύονται τι υπηρεσίε που ασχολούνται με την ασφάλεια τροφίμων, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι Ευρωπαίοι πολίτε πιστεύουν επίση ότι οι δημόσιε αρχέ κάνουν πολύ καλή δουλειά ενημερώνοντα το κοινό όσον αφορά του κινδύνου από τα τρόφιμα. Και αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόοδο σε σχέση με το 2005. Η δεύτερη μελέτη στην οποία αναφέρθηκα ολοκληρώθηκε στι αρχέ τη χρονιά αυτή και αξιολογεί πώ ε, αντιλαμβάνεται ο κόσμο την ΕΦΣΑ και πώς την ε, αξιολογούν Ιδίω οι εταίροι τη, οι διάφοροι φορεί, ε, μεταξύ άλλων ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οι εθνικέ υπηρεσίε ασφάλεια τροφίμων, οι εθνικοί οργανισμοί διαχείριση κινδύνου, οι επιστήμονε, τα μέσα ενημέρωση κλπ. Αντιλαμβάνονται λοιπόν όλη αυτή την έσφα σαν ένα ανοιχτό οργανισμό και διαφανή, ο οποίος παράγει πολύ σημαντικό έργο. Είμαστε δηλαδή για αυτούς ένας οργανισμός ο οποίος και παγιώνει αλλά και προσφέρει πραγματογνωμοσύνη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης δημιουργεί και συνέργειες μεταξύ των Εθνικών Υπηρεσιών Ασφάλειας Τροφίμων. Αναγνωρίζεται σαν ένας έμπιστος εταίρος που συνεισφέρει και στη διαχείριση, μάλλον στην αξιολόγηση του κινδύνου σε διεθνές επίπεδο. Έχουμε όλο και περισσότερες αιτήσει και όλο περισσότερες εντολές αναλαμβάνει η ΕΦΣΑ όπως ε, φαίνεται και εμείς προσπαθούμε να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματά μας όσον ε, αφορά την ασφάλεια τροφίμων όσο γίνεται περισσότερο ευρέως. Αναγνωρίζετε επίσης ότι η αξιολόγηση κινδύνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αυξηθεί χάρη στην οικονομική στήριξη που μας έχουν προσφέρει τα ευρωπαϊκά ε, θεσμικά όργανα. Είναι πολύ σημαντικό να διακρίνουμε την αξιολόγηση κινδύνου από τη διαχείριση κινδύνου. Είναι πολύ βασικό ε, να στοχεύουμε την ε, επιστημονική γνώση. Όσα απάντησαν στα ερωτηματολόγια μας, λένε ότι δεν θα έπρεπε να πάμε πίσω στην περίοδο που δεν υπήρχε η ΕΦΣΑ καθόλου. Παρ' όλα αυτά δεν εφησυχάζουμε, ξέρουμε ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, γιατί πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να αντιμετωπίζουμε με διαφάνεια ε, τα διάφορα θέματα, να είμαστε ανοιχτοί όπως σας είπα και να ε, παράγουμε ανακοινώσεις λιγότερο τεχνικές. Και αυτό θα κάνουμε το 2011 και μετά. Αν δούμε λοιπόν τι έχουμε πετύχει τα τελευταία 8 χρόνια, μπορούμε να πούμε ότι γενικά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλειας Τροφίμων έχει προσφέρει πολλά και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ιδρυτών ε, πατέρων και μητέρων, γιατί όχι. Η Ευρώπη λοιπόν έχει πετύχει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τα θέματα υγείας που έχουν να κάνουν με τα τρόφιμα. Σαλμονέλα, σπογγώδησε κεφαλοπάθεια των βοηδών, ε, χημικές ουσίες. Η ΕΦΣΑ έχει συνεισφέρει θετικά στα επιτεύγματα αυτά. Επιπλέον, για να φέρει σε πέρα στην αποστολή της, η ΕΦΣΑ έχει προσαρμοστεί με ρυθμιστικές αλλαγές όσον αφορά την ε, διαχείριση κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα εργασίας της ΕΦΣΑ έχει εξελιχθεί, έχει αλλάξει και όσον αφορά το εύρος του και όσον αφορά τη φύση του. Αν δούμε καθαρά ποσοτικά τα πράγματα, θα έλεγα ότι η παραγωγή έργου μας έχει επιταχυνθεί πολύ για να αντιμετωπίσουμε τα όλο και αυξανόμενα αιτήματα που λαμβάνουμε. Αν συγκρίνουμε, το 2007 είχαμε 220 αιτήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2009 αυξήθηκαν στα 360 και το 2010 είχαμε 900. 900 ερωτήσεις από την Κομισιόν. Αυτή η σημαντική αύξηση όσον αφορά την παραγωγή έργου πάνω από 600 ήδη φέτος για να αντιμετωπίσουμε το αίτημα έχει προχωρήσει χάρη στο συνδυασμό και οικονομικών πόρων αλλά και προσωπικού. Έχουμε καταφέρει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να έχουμε την στήριξη από επιστήμονες, από ειδικού και βέβαια εκτός των άλλων έχουμε και την προσπάθεια που κάνει το ίδιο το προσωπικό της ΕΦΣΑ που είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένο στο έργο του. Οι εξελίξει όσον αφορά το ρυθμιτικό πλαίσιο λοιπόν από το 2002 και μετά έχουν συνεισφέρει πολύ στο αποτέλεσμα για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε και να απαντάμε σε όσο γίνεται περισσότερες απαντήσεις. Με θέματα όπως είναι τα εντομοκτώνα, όπως είναι οι ζωοτροφές, τα τρόφιμα φυσικά για ανθρώπινη κατανάλωση, ε, οι ουσίες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα κλπ. Θα ήταν δύσκολο να τα καταφέρουμε όλα αυτά πριν από 8 χρόνια δεν θα είχαμε φανταστεί ποτέ ότι το 70% του επιστημονικού μας έργου θα είχε να κάνει με αιτήσει ε, στις οποίες πηγαίνει το 40% των πόρων μας. Έτσι λοιπόν το πρόγραμμα εργασίας της ΕΦΣΑ μοιάζει πάρα πολύ με το πρόγραμμα εργασίας άλλων οργανισμών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων, η ΕΚΑ. Η φύση του έργου μας έχει επίσης εξελιχθεί για να ανταποκριθούμε σε αλλαγές στο νομοθετικό επίπεδο. Η ΕΦΣΑ λοιπόν δεν αξιολογεί μόνο τους κινδύνους για τους ανθρώπους και τα ζώα όσον αφορά την υγεία, αλλά αξιολογεί και τη ζημιά στο περιβάλλον. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε τις επιπτώσεις των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε και το περιβάλλον και να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής τροφικής αλυσίδας. Επιπλέον, ε, μας ζητείται όλο και περισσότερο να αξιολογούμε όχι μόνο κινδύνους, αλλά και την αποτελεσματικότητα ή τα ωφέλη για την υγεία ή για το περιβάλλον. Και αυτό κάνουμε όσον αφορά τα εντομοκτώνα, για παράδειγμα. Επίση, έχουμε επενδύσει πολύ στην συλλογή δεδομένων για να μπορούμε την αξιολόγηση κινδύνου να την κάνουμε επάνω σε στέρεες βάσεις. Ο έλεγχος είναι πολύ βασικός για να προστατεύουμε τους καταναλωτές και το περιβάλλον. Η ανακατανομή των πόρων τώρα που χρειάστηκε να θέσουμε σε εφαρμογή ανταποκρίνεται στο γεγονό ότι έχουν αυξηθεί οι αιτήσει που λαμβάνουμε. Άρα λοιπόν έπρεπε να θέσουμε διάφορα σημαντικά ερωτήματα στου εαυτού μα. Πρώτα απ' όλα, πώ μπορούμε να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε ε, το θέμα των κινδύνων στην υγεία από χημικού παράγοντε, βιολογικού παράγοντε ή θέματα που έχουν να κάνουν με τη διατροφή, ενώ συγχρόνως με την δουλειά μα πρέπει και να υποστηρίξουμε την στρατηγική 2020 ε, που αποτελεί να βαρχίδα για την Ευρώπη όσον αφορά την καινοτομία. Θα σας πω λοιπόν πώς προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την διπλή πρόκληση. Με τέσσερα βήματα. Πρώτον, έχουμε το σύστημα του πάνελ που πιστεύουμε ότι είναι αξιόλογο και ότι προσφέρει αποτελέσματα όπως θα θέλαμε. Όμως, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είναι και βιώσιμο. Έχουμε, όπως σας είπα, όλο και περισσότερες αιτήσει. Γι' αυτό ένα μεγάλο ποσοστό των εμπειρογνωμών μα ασχολείται με τις αξιολογήσεις ρουτίνας. Όμω, εξαιτία τη τρέχουσα οικονομική κατάσταση, είναι όλο και πιο δύσκολο για του εθνικού εμπειρογνώμονε ε, να συμμετέχουν στο έργο μα. Για να μπορούμε λοιπόν να γίνουμε πιο ελκυστικοί για σπουδαίους εμπειρογνώμονε. πρέπει να εξυγχρονίσουμε τον ρόλο των πάνελ. Γι' αυτό και προτείνουμε στο μέλλον να επικεντρωθούμε εκεί όπου η πραγματογνωμοσύνη μπορεί να έχει και μεγαλύτερα αποτελέσματα. Να ασχοληθούμε δηλαδή τα πάνελ αυτά, να ασχολούνται με πιο σημαντικά θέματα και να αναπτύξουμε μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση κινδύνου, χωρίς βέβαια να πληγεί η ποιότητα του έργου μας. Δεύτερον, σαν αποτέλεσμα των αλλαγών αυτών, στο που δίνουμε την έμφαση στο έργο των εμπειρογνωμόνων, η ΕΦΣΑ θέλει να αυξήσει τον αριθμό του επιστημονικού προσωπικού που ασχολείται με την επεξεργασία των αιτήσεων. Έχουμε ήδη εφαρμόσει ένα τέτοιο μοντέλο στον τομέα των εντομοκτών σε συνεργασία με εθνικές υπηρεσίες ε, αξιολόγησης κινδύνου, όπως γίνεται και στην EMA. Είναι πολύ βασικό επίσης να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον όγκο των αιτήσεων και αυτό μπορούμε να το κάνουμε αν από πριν μπορούμε να εκτιμήσουμε πόσες αιτήσει θα έχουμε. Η επιστημονική κοινότητα σκέφτεται πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε καλύτερα τις συμβάσεις που ετησίως προσφέρουμε. Είχαμε 1 εκατομμύριο το 2007 ευρώ, 1 εκατομμύριο ευρώ, με 8 εκατομμύριο το 2010. Περιορισμοί όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες ολόκληρη την Ευρώπη μας αναγκάζει, την ΕΦΣΑ δηλαδή, να συνεργάζεται στενά με τα κράτη-μέλη. Πρέπει να αναπτύξουμε παρετέρω τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη, λοιπόν, και με τα κράτη-μέλη συμφωνήσαμε ότι στην εργασία μας θα επικεντρωθούμε σε ένα συγκεκριμένο αριθμό εθνικών οργάνων, που είναι τα κέντρα αριστείας, που επενδύουν σε συγκεκριμένους τομείς πραγματογνωμοσύνης. Θα είναι μια νέα προσέγγιση αυτή, από την οποία αμοιβαία θα υποφεληθούν και η ΕΦΣΑ και τα κράτη-μέλη. Η ΕΦΣΑ, διότι θα μπορέσει να βοηθήσει αποτελεσματικά με το έργο της και να ε, πολλαπλασιάσει ουσιαστικά τις επιτυχίες και συγχρόνως στηρίζουμε και τις δυνατότητες που έχουν τα κράτη-μέλη. Αλλά το επίπεδο επενδύσεων 8 εκατομμυρίων θα πρέπει να αυξηθεί. Τέταρτον, ανακοινώσεις όσον αφορά το κίνδυνο. Είναι κάτι που γίνεται και από την πλευρά των εκείνων που αξιολογούν τον κίνδυνο, αλλά και εκείνων που διαχειρίζουν τον κίνδυνο. Έχουμε αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες μέχρι τώρα για μια νέα στρατηγική 2010-2013. Θέλουμε να βασιζόμαστε και τις ανακοινώσεις μας στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Θα αναπτύξουμε μια πιο καταθέμα προσέγγιση όσον αφορά τις δραστηριότητές μας αυτές. Παρόλο που κάθε επιστημονικό μας αποτέλεσμα το δημοσιοποιούμε και το δημοσιεύουμε, θα φροντίσουμε να είμαστε πιο δραστήριοι στις ανακοινώσεις μας, εκεί όπου μπορούμε να προσφέρουμε και αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ακούσαμε τα βασικά μηνύματα και τώρα θα περάσουμε στις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση από την Πιλάρ Αγιούζο, από το ΕΛΚ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συγγνώμη για τη φωνή μου, λέει η ομιλήτρια, που είναι βραχνιασμένη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τζεσλέν, για τα επιστημονικά αποτελέσματα και την ανακοίνωσή τους προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά και άλλα όργανα και υπηρεσίες. Είναι μεγάλη ευθύνη. Χθε λέγαμε ότι πολλές μελέτες ίσως δεν είναι ανεξάρτητες από τη βιομηχανία. Μερικές φορές ε, μιλούσαμε τότε για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, έτσι. Και θυμήθηκα ότι το γιο μου όταν παίζει ποδόσφαιρο, όταν χάνει η ομάδα του, φταίει ο διαιτητής. Όταν κερδίζει η ομάδα του, είναι δικό του το κέρδος. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρό να έχουμε μία ε, επιστημονική επιτροπή, αλλά έχετε συγχρόνως και 10 επιμέρους επιστημονικές ομάδες. Πώς γίνεται το έργο σας εκεί, οι ομάδες αυτές είναι πραγματικά ανεξάρτητες από τη βιομηχανία. Η ΕΦΣΑ έχει επιστήμονες οι οποίοι θα πρέπει να είναι εντελώ ε, ανεξάρτητοι. Αυτά που άκουσα εδώ χτες που κατηγορήθηκαν επιστήμονες ότι έχουν άμεση σύνδεση με τη βιομηχανία μου φάνηκαν πολύ ανησυχητικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είπατε, εμείς στηριζόμαστε σε εξωτερικές επιστημονικές ε, συμβουλές. Γι' αυτό από τις αρχές την δημιουργία της ΕΦΣΑ δημιουργήσαμε μια, μια πολιτική εξωτερικών συμβουλών, αν θέλετε. Έχουμε ενδυναμώσει την πολιτική αυτή το 2007 και στηριζόμαστε σε έξι πυλώνες. Όπως είπατε, ε, ο πρώτος πυλώνας είναι η επιλογή των εμπειρογνωμόνων και τα κριτήρια είναι διάφανα επιλογής τους και είμαστε σίγουροι ότι έχουν υψηλό βαθμό επιστημονικών ε, γνώσεων, έχουν εμπειρία για επιστημονικές αξιολογήσεις και προφανώς δεν έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα. Επίσης, εργάζονται σε πάνελ και σε επιτροπές και σε ομάδες εργασίας, δηλαδή ε, λειτουργούν συλλογικά. Δεν στηρίζεται ποτέ η ΕΦΣΑ στην μεμονωμένη παροχή συμβουλών και στα 20 κάτι μέλη του πάνελ στηριζόμαστε. Επίσης, κάθε εμπειρογνώμονας πρέπει να δηλώσει όλα του τα συμφέροντα, σε αυτή την ετήσια δήλωση συμφερόντων που δημοσιεύεται νηστό τοπό μας και πριν από κάθε συνεδρίαση, ανάλογα με το περιεχόμενο της ημερήσιας διάταξης, κάνει μία δήλωση συμφερόντων η οποία ελέγχεται από το προσωπικό μας μετά την μελέτη αυτού του, αυτής της δήλωσης ο εμπειρογνώμονας μπορεί να μην πάρει μέρος στην συνεδρίαση ούτε σαν μέλος ούτε σαν εισηγητής ούτε σαν πρόεδρος. Επίσης έχουμε δημιουργήσει μια πολιτική σύμφωνα με την οποία εάν κάποιος εμπειρογνώμονας δεν κάνει την δήλωση αυτή έχουμε τα κατάλληλα μέτρα. Πρόσθετη ερώτηση, όχι, η Dagmar Για να αρχίσει το χρονόμετρο, περιμένω. Μάλιστα. Μηδεν είστε το παρακαλώ. Πολύ σύντομα. Κυρία Γκισλά Λανοέλ, για την επιστημονική αριστεία. Πώς νομίζετε ότι μπορείτε να βελτιώσετε την επιστημονική αριστεία λαμβάνοντας υπόψη και την αρχή της προφύλαξης που είναι μια βασική αρχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα αυξήσετε την εμπιστοσύνη στις γνωμοδοτήσεις της ΕΦΣΑ και των επιστημόνων. Με όλα τα μέσα που έχετε λάβει σίγουρα δεν φτάνει το βαθμό που θα θέλαμε να υπάρχει τέτοιου είδου ε, αξιοπιστία. Και είπατε σχετικά με το σύστημα των πάνελ ότι μπορεί να αλλάξει. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει το σύστημα τη ΕΦΣΑ. Δεν ξέρω για το σύστημα των πάνελ αν πρέπει να αλλάξει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με την αλλαγή δομή που θέλετε, τι θα κάνετε αν δεν έχετε τα χρήματα και το προσωπικό που χρειάζεστε. Αν παράλληλα θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη να αλλάξετε τα πράγματα. Και ένα τελευταίο σημείο για την πολυπλοκότητα των επιστημονικών απόψεων για να λαμβάνουν υπόψη και τις κοινωνικές ανάγκες. Ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις σε ένα λεπτό. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι η ποιότητα είναι ε, υψίστης σημασία, διότι δεν είναι απλώς και μόνο ανεξάρτητες επιστημονικές ε, συμβουλές ή δεδομένα. Θέλουμε να έχουμε και την ε, βέλτιστη δυνατή ποιότητα. Επίσης δεν, ε, είμαστε, δεν συγκεντρωνόμαστε μόνο στην, ε, στην Ευρώπη αλλά και στο ιστορικό για την αξιολόγηση των κινδύνων. Επίσης έχουμε αναπτύξει στην ΕΦΣΑ ε, τεχνικές συλλογής δεδομένων και πληροφοριών. Επίσης ελέγχουμε και τις αβεβαιότητες. αυτή είναι μία μέθοδος που εφαρμόσουμε στην ΕΦΣΑ έτσι ώστε να αξιολογούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο του κινδύνου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την αρχή της προφύλαξης. Επίσης ε, στο οργανώμα γραμμά ε, κάθε χρόνο για το οργανόγραμμά μας ε, ελέγχουμε 800 αιτήσει κάθε χρόνο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πρόβλημα δεν είναι το οργανόγραμμα μόνο, αλλά συνεργαζόμαστε και με έναν εξωτερικό σύμβουλο έτσι ώστε να βελτιώσουμε τα μεταρρυθματικότητα της εργασίας μας. Επίσης, οι κοινωνικές ανάγκες. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι θα πρέπει να έχουμε την ευέλτιστη καλή επιστημονική συμβουλή, μέσα στα πλαίσια όμως των ε, εντολών που έχουμε πάρει, που είναι η δημόσια υγεία, η ανθρώπινη υγεία, η υγεία των ζώων, των φυτών κτλ. Η πρέπει να κάνουμε και περιβαλλοντικές ε, ε, αξιολογήσεις των κινδύνων. Ε, πρέπει επίσης να αξιολογήσουμε και την αποτελεσματικότητα στην βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. Επομένως, μπορούμε Μπορούμε να διευρύνουμε τι αρμοδιότητέ μας όμως μόνο μέσα στα πλαίσια του κανονιστικού πλαισίου. Άλλες ερωτήσεις δεν ζήτησα να διευρυνθεί η... Ε, το, η αρμο, να, να βρεθεί το πλαίσιο αρμοδιοτήτων ε, της ΕΦΣΑ, αλλά απλώς να διευρυνθεί το πλαίσιο λειτουργίας των επιστημόνων που δουλεύουν για την, ε, για την ΕΦΣΑ, διότι ε, πραγματικά δεν κάνουν αυτό το οποίο τους ζητάμε. Πώς μπορείτε να τους εκπαιδεύσετε. Πρέπει να τους επαναλάβετε, να τα ξέρουν πώς ε, πρέπει να γίνουν ε, οι, οι απαραίτητες αλλαγές στην ΕΦΣΑ χωρίς αναγκαστικά να πάρετε ούτε περισσότερα χρήματα ούτε περισσότερο προσωπικό. Κοιτάξτε, έχουμε καταβάλει πολλές προσπάθειες ε, για να βελτιώσουμε την διαφάνεια ε, των επιστημονικών μας μεθόδων. Ε, μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα σε κάποιους τομείς ίσως, όπου σίγουρα στους γενετικά ας πούμε τροποποιημένους οργανισμούς οι συμβουλές της ΕΦΣΑ, οι οι απόψει τη ΕΦΣΑ δεν είναι οι, οι, Άρα εκεί μπορούμε να βελτιωθούμε. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι αρμοδιότητες της, της ΕΦΣΑ περιορίζονται μόνο στην αξιολόγηση των κινδύνων. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παραπάνω, διότι αλλιώς θα, θέσουμε σε κίνδυνο τον, τον διαχωρισμό της αξιολόγησης του κινδύνου και της διαχείρισης του κινδύνου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ερώτησή μου προ την κυρία Διευθύντρια θα είναι προ την ίδια κατεύθυνση με αυτή που έθεσε η κυρία Αγιούζο. Μα είπατε ότι έχετε κάνει πολλέ προσπάθειε και βεβαίω σα το αναγνωρίζουμε, αλλά έχω μια πολύ απλή ερώτηση. Σε αυτή τη δεύτερη θητεία έχετε την πρόθεση ε, να ε, ε, συμβαδίζουν οι πράξεις σας με αυτά τα οποία μας είπατε. Το Ηλσι, το Διεθνές Ινστιτούτο για τις επιστήμες οι φυσικές επιστήμες ε, θα συνεχίσει το έργο του. Σκέφτομαι τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, τον κύριο Κέιπερ και τον κύριο Κρίτερ. Οι προτάσεις ε, του ΙΛΣΙ, του Ινστιτούτου αυτού, σε μεγάλο μέρος επαναλαμβάνονται μέσα στις κατευθυντήριες γραμμές. Μήπως πρέπει να επανεξετάσετε το πάνελ για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και να περάσετε από την αναζήτηση της συνένεσης, που δεν έχει μεγάλο νόημα παρά μόνο ότι εμποδίζει τις κριτικές, σε μια πραγματική αντιπαράθεση που θα δίνει τη δυνατότητα και σε απόψεις μειοψηφία και σε επιστημονική στάση. Ευχαριστούμε. Απάντηση. Όπως είπα, το ενδιαφέρον ε, των ε, ε, τα διάφορα συμφέροντα των εμπειρογνωμόνων που είναι μέλη των πάνελ ελέγχονται με βάση πολύ διαφανή κριτήρια που είναι ανοιχτά προς όλους. Και είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι η ΕΦΣΑ στο έργο της λαμβάνει υπόψη όλες τις ε, ορθές και χρήσιμες επιστημονικές πληροφορίες από όπου και αν προέρχονται. μπορεί να προέρχονται από επιστημονική βιβλιογραφία, από τους φακέλους που υποβάλλει ο ετών, μερικές φορές από κάποιες ε, ε, συνεισφορές από φορείς που χρηματοδοτούνται από τον κλάδο, από τη βιομηχανία. Εμείς θέλουμε να είναι ορθές επιστημονικές γνώμες. Όταν μιλάμε για ανεξαρτησία της ΕΦΣΑ, φροντίζουμε να μην ξεχνάμε το γεγονός ότι οφείλουμε να είναι σωστό το επιστημονικό μας αποτέλεσμα. Οι συμβουλές μας πρέπει να είναι και ανεξάρτητες βέβαια και αυτό το έχουμε κατά νου. Αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζει η επιστημονική κοινότητα, η κοινότητα που κάνει την αξιολόγηση κινδύνου και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπη. Και θεωρείται ότι είναι πολύ καλή αξιολόγηση κινδύνου που κάνουμε. Σε σχέση με αυτό που είπατε κυρία Λεπάζ, θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό το να έχουμε ανοιχτή συζήτηση με αντιπαράθεση απόψεων, με εμπειρογνώμονες που έχουν διαφορετικές απόψεις. Στην ομάδα εργασίας θέλουμε όλο και περισσότερο να υπάρχει δυνατότητα να καλούμε και κάποιους εμπειρογνώμονες σε ακρόαση, δηλαδή κάποιους εμπειρογνώμονες που ενδέχεται να θεωρούμε ότι έχουν και σύγκρουση συμφερόντων, μπορεί να προέρχονται από τη βιομηχανία ή από μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αρκεί να έρχονται στην ακρόαση αυτή με τις κατάλληλες πληροφορίες και απόψεις ε, για να τους ακούσουμε. Και όταν υπάρχει αντιπαράθεση, όταν γίνεται μια συζήτηση για ένα επιστημονικό θέμα, περιλαμβάνουμε τη συζήτηση αυτή και στο επιστημονικό έργο της ΕΦΣΑ όταν γίνεται κάτι στην κοινή γνώμη γενικότερα. Κύριε Λεπάζ, ε, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν απαντήσατε στην πολύ συγκεκριμένη μου ερώτηση για το Ινστιτούτο Ήλση. Ο κύριος Σκουιπέρ είναι υπεύθυνο του πάνελ για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, δηλαδή κάποιος που έχει μεγάλη αρμοδιότητα και θα ήθελα μια επακριβή απάντηση στην ερώτησή μου, παρακαλώ. αν δεν κάνω λάθος, οι δραστηριότητες στις οποίες αναφέρεστε έχουν σχέση με το ότι πριν από λίγα χρόνια προέκυψε ένα έγγραφο για την αξιολόγηση κινδύνου και τη σχετική μεθοδολογία για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Αυτό ήταν το θέμα και έρευνας που χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας πρόγραμμα δηλαδή με δημόσια χρηματοδότηση και ο κύριος Σκόιπερ όπως και άλλοι εμπειρογνώμονες ασχολήθηκαν με αυτό το πρόγραμμα. Αυτή τη δραστηριότητα τη θεωρούμε σίγουρα χρήσιμη προς τη δουλειά του πάνελ και το επιστημονικό πάνελ της ΕΦΣΑ δεν ε, ευλόγησε ή δεν ενέκρινε αυτό το έγγραφο. Υπήρξαν και πολλές άλλες συνεισφορές λαμβάνοντας, ε, που λήφθηκαν υπόψη από τις δραστηριότητες του πάνελ όταν ε, επεξεργάστηκε τη μεθοδολογία. Ευχαριστώ πολύ. Μπαρτ Ευχαριστώ. Θέλω να επιμείνω και εγώ στην ερώτηση της κυρίας Αγιούσο και της κυρίας Λεπάς Και εγώ, μέσω του Ευρωβαρομέτρου, έχω την εντύπωση ότι θεωρείται πολύ σημαντικό θέμα την ανεξαρτησία. Και πράγματι, ο διευθυντή ενό τέτοιου οργανισμού όπω είναι η ΕΦΣΑ πρέπει να φροντίσει να μην υπάρχει σύνδεση με τη βιομηχανία. Όμω για το θέμα ακριβώ αυτό τη ανεξαρτησία των ε, επιστημόνων σας, από το 2007 φροντίσατε να υπάρχουν έξι κατευθυντήριες γραμμές. Στη θεωρία πολύ ωραίο αυτό. Στην πράξη όμως, πόσες φορές έχετε διαπιστώσει ότι ένας ε, εμπορογνώμων, ένας εμπειρογνώμων τελικά έδωσε κάποια στοιχεία ή είδατε ότι δεν ήταν απόλυτα ανεξάρτητος. Πότε τέθηκε σε κίνδυνο η ανεξαρτησία αυτή δηλαδή των πάνελ σας. Ποια είναι η πραγματικότητα σε σχέση με αυτήν τη θεωρία. Μπορείτε να μας διαφωτίσετε περισσότερο σε αυτό. So, um, Όπως είπα, έχουμε καθορίσει με σαφήνεια στην πολιτική μας όσον αφορά ε, την επικάλυψη συμφερόντων Ποιες είναι οι διαδικασίες σύγκρουση συμφερόντων. Λέμε τι είναι συμφέρον, τι είναι σύγκρουση συμφερόντων και βάσει αυτού καθορίζουμε την πολιτική μας που φροντίζουμε και να εφορμόζουμε στην καθημερινή μας δουλειά. Τώρα τα κριτήρια σε σχέση με άλλους οργανισμούς τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός Ευρώπης νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι για το ότι τα δικά μας τα κριτήρια είναι πολύ καλά. Η πολιτική μας δηλαδή είναι στεναρή. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να εφαρμόσετε τα κριτήρια για να δείτε αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ή όχι. Και για τα κριτήρια ευχαρίστω να το συζητήσω και μαζί σας. Αλλά επιπλέον μπορώ να σας πω ότι μετά από τρία χρόνια εφαρμογής της πολιτικής μας αυτής και ακριβώ επειδή έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό και με την αντιπροσωπεία σας που ήρθε στην Πάρμα, συζητήσαμε το ότι οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι των επιστημονικών επιτροπών και εμπειρογνώμονε ε, είναι πιο υπεύθυνοι από τους άλλους, γιατί είναι περισσότερο ορατοί και ίσως θα πρέπει να, είναι, να είμαστε πιο αυστηροί. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε και νέα μέσα, ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων που έχουμε ορίσει, για να αποφύγουμε δυνητικά κάποια σύγκρουση συμφερόντων όταν πρόκειται για τέτοιες θέσεις. Και έχουμε ήδη υιοθετήσει μέτρα και του χρόνου και μετά όταν θα έχουμε τα ονόματα για όλα τα πάνελ θα φροντίσουμε να εφαρμοστούν αυτοί οι κανόνες. Ο κύριος Στάση. Ευχαριστώ για την απάντησή σα, αλλά η συγκεκριμένη μου ερώτηση είναι, τα τελευταία τρία χρόνια, τέλο πάντων όσοι είσαστε εσεί εκτελεστικό διευθυντή, υπήρξαν κάποιοι εμπειρογνώμονε εξωτερικοί οι οποίοι να μην τήρησαν του κανόνε ή μέσα από το screening που εφαρμόζεται να φάνηκε ότι υπήρξε κάποια σύγκρουση συμφερόντων ή μπορέσατε να προλάβετε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις υπήρξαν συμφέροντα στη βιομηχανία, στην πραγματικότητα δηλαδή. Είχατε τέτοιες περιπτώσεις. Yes, Ναι, κάθε εβδομάδα έχουμε εμπειρογνώμονες που τους αποκλείουμε από κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες είτε δεν μπορούν να προεδρεύσουν, είτε δεν μπορούν να είναι εισηγητές, είτε συντάκτες. Κάθε εβδομάδα. Συνηθίζεται για να τηρηθεί η ανεξαρτησία. Δεν είναι δηλαδή κάτι έκτακτο. Μάλιστα υπάρχει και περίπτωση όπου δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι ένας εμπειρογνώμονας παρέλειψε να δηλώσει κάποια συμφέροντα. Δύο φορές. Και ξεκινήσαμε διαδικασία επάυσης των εμπειρογνωμόνων αυτών. Και όχι μόνο αυτών, ελέγξαμε και το επιστημονικό έργο για να διασφαλίσουμε ότι η επιρροή του πυρογνώμων αυτού δεν ήταν τέτοια που να μπορούσε να θέσει υπομφισβήτηση το έργο μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση για την κλωνοποίηση και ιδιαίτερα το τι κάνετε για τα πρότυπα που αφορούν τα ιδιατροφή στα κράτη-μέλη και πώς ε, γίνεται η ανταλλαγή πληροφοριών και συμβουλών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Παρασκευή, ακούσαμε ότι είναι ασφαλές ε, το να τρώει κανείς κλωνοποιημένο κρέας. Αυτό συμπληκτεί και με τις απόψει του φορέα σα, ότι δεν υπάρχει ένδειξη ότι υπάρχει κάποια διαφορά αλλά δεν είναι ακριβώς η ίδια η απόχρωση, δεν είναι τόσο ε, καταφατική αυτή η απάντηση και δεν δίνει συμβουλές ε, προς τους καταναλωτές. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πώς οργανώνετε τι επαφές σα με τα κράτη-μέλη για τέτοια θέματα και πώς συμπεριλαμβάνετε τις αποφάσεις των κρατών μελών και την πληροφόρηση από τα κράτη-μέλη στη δική σας ε, πληροφόρηση και αν ε, προβλέπετε κάποια χωριστή νομοθεσία για τα κλωνοποιημένα ζώα. Σας ευχαριστώ. Αν πάρουμε το παράδειγμα της κλωνοποίησης, Χρησιμοποιούμε πολλούς τρόπους συνεργασίας με τα κράτη-μέλη. Καταρχήν, όταν μας ζητήθηκε από την Επιτροπή να εκδώσουμε μια επιστημονική συμβουλή για το θέμα, συνεννοηθήκαμε με τους ε, εμπειρογνώμες με τους οποίους είμαστε σε επαφή σε όλα τα κράτη-μέλη για να πάρουμε όλα τα δεδομένα και για να ορίσουμε τους σωστούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα αποτελούσαν την ομάδα εργασίας για το θέμα αυτό. Και αυτό είναι ουσιαστική σημασία γιατί γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν τόσο πολλά στοιχεία και τόσο πολλές πληροφορίες, επομένως ήταν κέρια σημασία να συλλέξουμε όσα υπήρχαν διαθέσιμα. Πρέπει να πω ότι η δήλωση που έγινε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων υποστηρίζεται από τις επιστημονικές συμβουλές της ΕΦΣΑ δήλωσαν ότι δεν έχουν διαφωνία με αυτά τα οποία είπαμε για την ασφάλεια, για την διαφορά δηλαδή μεταξύ γάλακτος ή κρέατος που προκύπτουν από κλωνοποιημένα ζώα ή τους απογόνους τους. Ε, Παρ' όλα αυτά υπάρχει ε, μια επιφύλαξη για την ε, υγεία και την ε, ευζοία των ζώων, πράγμα το οποίο είναι και αυτό μέσα στις αρμοδιότητές μας. Υπάρχουν αρκετές αβεβαιότητες στον τομέα αυτό και γι' αυτό συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το θέμα πάρα πολύ στενά. Έχουμε ήδη ενημερώσει την επικαιροποίηση την επιστημονική μας δήλωση και παρακολουθούμε και την ανάπτυξη κάποιων βασικών ερευνητικών προγραμμάτων στα κράτη-μέλη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις αβεβαιότητες και το κενό γνώσεων που υπάρχουν σε αυτό τον τομέα. Δεν μπορώ να σχολιάσω επίσης για την νομοθεσία γιατί δεν είναι τμήμα της δικής μας αρμοδιότητας. Δεν αναμένεται από εμά να σχολιάσουμε το αν πρέπει να υπάρχει χωρίς την νομοθεσία για την κλωνοποίηση ή όχι. Σας ευχαριστώ. Ναι, νομίζω ότι ε, με αυτά που είπατε δείξατε αυτό που ήθελα να πω και εγώ, ότι υπάρχει πολιτιστική διαφορά στις γνωμοδοτήσεις. Μπορεί να πρόκειται για επιστημονικά δεδομένα, αλλά η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να, να πει ότι ε, ολοκληρώθηκε η συζήτηση, είναι ασφαλές το κρέας από κλωνοποιημένα ζώα. Εσείς λέτε ότι εμείς συνεχίζουμε τις έρευνες και μπορεί να μην σας δώσουμε καθόλου απάντηση. Δεν λέω ποιο έχει δίκιο και άδικο, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή είναι και καθήκον σας κάποια στιγμή να δίνετε μια απάντηση στους καταναλωτές. Ναι, νομίζω ότι δίνουμε απάντηση όταν λέμε ότι αυτή είναι η κατάσταση των πραγμάτων και πρέπει να συνεχίσουμε τη στενή παρακολούθηση. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την κλωνοποίηση, αλλά για όλε τι επιστημονικέ συμβουλέ που δίνετε. Ποτέ δεν θα ακούσετε να σα πούμε ότι είναι ασφαλέ, τελεία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμεί, ω σοβαρό οργανισμό, πρέπει να πούμε ότι η επιστήμη εξελίσσεται, αλλάζει καθημερινά και αυτό το οποίο σήμερα είναι αλήθεια μπορεί αύριο να αποδειχθεί ασφαλμένο. Γι' αυτό πάντοτε πρέπει να είμαστε μετριοπαθεί και αυτό προσπάθησα να σα πω ότι δεν είναι εύκολο να ε, περνάει η επικοινωνία για τα ευρήματά μας. Ευχαριστώ. Κάτι καλλιόκα. Ευχαριστώ. <clears throat> Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Είσαστε η μόνη υποψήφια. Υπήρξε ανοιχτή διαδικασία υποψηφιότητων. Πώς γίνεται που εσείς είσαστε η υποψήφια. Γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες, είναι δύσκολη η δουλειά στην ΕΦΣΑ, υπερβολικός φόρτος, ή οι οικονομικά μέσα δεν είναι αρκετά και γι' αυτό δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφοι που να ενδιαφέρονται. Μήπως πρέπει κάτι να αλλάξει για να υπάρχουν ε, περισσότεροι πόροι. Είναι αυτή η δυσκολία. Um, thank you Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Η ακρόαση αυτή αποτελεί μέρος μια διαδικασίας που περιγράφεται ε, με λεπτομέρειες στα ιδρυτικά μας κείμενα που λέει ότι ο εκτελεστικός διευθυντής μπορεί μία φορά να ζητήσει την επανεκλογή του. Γι' αυτό και υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος που είμαι εγώ. Αλλιώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προκυρήσει διαγωνισμό. Έτσι έχει η διαδικασία. Θέλω εδώ να σας πω ότι πράγματι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε παραπάνω φόρτο εργασίας, ότι είμαστε στο τέλος ε, μιας περίοδου της ΕΦΣΑ. Είμαστε περήφανοι βέβαια και ευχαριστημένοι που έχουμε παραπάνω δουλειά, γιατί αυτό δείχνει ότι μας εμπιστεύεστε. Είναι αλήθεια όμως ότι μεταξύ μας συζητάμε το ότι η ΕΦΣΑ πρέπει να έχει τις δυνατότητες να φέρει σε πέρα στην αποστολή της. Είτε πρόκειται για τα χημικά, είτε πρόκειται για βιολογικούς παράγοντες, τα τρόφιμα, είτε πρόκειται για κάτι άλλο. Υπάρχει η δουλειά ροτίνας, αλλά υπάρχει και έκτακτη δουλειά. Όλα είναι σημαντικά. Ο λόγος ύπαρξης της ΕΦΣΑ, μην ξεχνάμε, είναι η προστασία των καταναλωτών από ασθένειες όπως είναι η σπογγόδης ε, κεφαλοπάθεια. Τώρα ασχολούμαστε και με τα τρόφιμα. Πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν η ΕΦΣΑ να μπορεί να κάνει και τα δύο στο μέλλον και να στηρίζει την βιώσιμη καινοτομία και να στηρίζει την αξιολόγηση κινδύνου από τα τρόφιμα. Και τα δύο θέλουμε να τα κάνουμε. Συμπληρωματική ερώτηση. Ναι, αλλά εγώ σας ρωτάω και για την χρηματοδότηση της ΕΦΣΑ. Μήπως πρέπει να ξανασκεφτείτε το σύστημα χρηματοδότησής σας. Τι θα κάνετε, τι σκέφτεστε γι' αυτό, πώς θα συνεργαστείτε ώστε να διασφαλίσετε την ε, επίτευξη του έργου της ΕΦΣΑ. Well, here I would say... Εδώ πρέπει να σας πω ότι πιστεύω πως βάσει το ράματος της ΕΦΣΑ μπορούμε να ζητήσουμε επιπλέον χρηματοδότηση. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν οικονομικές και δημοσιονομικές δυσκολίες επί του παρόντος. Γι' αυτό δεν θα έκανα έκκληση ούτε για παραπάνω πόρους στον προπολογισμό μας, ούτε για έκτακτη χρηματοδότηση. Όμως ζητούμε την δικιά σας στήριξη για να μπορούμε να προστατεύουμε τους καταναλωτές. Ο μόνος τρόπος για να έχουμε παραπάνω πόρους είναι να έχουμε ένα σύστημα επιπλέον χρημάτων για την κάποιο είδου τελών Υπάρχουν άλλοι οργανισμοί όπως η Υπηρεσία Φαρμάκων, ε, Χημικών που εφαρμόζει ένα τέτοιο σύστημα. Και όντως μπορούμε να το σκεφτούμε για να μπορούμε να διασφαλίσουμε πλήρως την ανεξαρτησία. E Σας ευχαριστώ πολύ να περάσουμε στο δεύτερο γύρο, η Ρενάτε Ζόμερ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Έχω μια ερώτηση για τον κανονισμό, για τους ισχυρισμούς για θέματα υγείας. Πρέπει να αξιολογήσει χιλιάδες ισχυρισμούς ε, υγείας, ε, περίπου 4.000 είπατε ε, και δεν ξέρω αν θα, χειριστείτε όλο τον κατάλογο παράλληλα. Μπορεί να γίνει ε, ε, η εξέταση όλων των ισχυρισμών μαζί ή θα δώσετε κάποια προτεραιότητα. Πώς θα κλιμακώσετε την εξέταση των ισχυρισμών. Το δεύτερο ερώτημά μου για την χρέωση τελών από την αίθουσα στο μέλλον. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα ισχύσει και για την αξιολόγηση των ισχυρισμών υγείας τι κάνει η ΕΦΣΑ για να λάβει υπόψη την κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επιβαρύνονται πάρα πολύ. Θα υπάρξει κάποια κλιμάκωση στα τέλη που επιβάλλονται. Θα είναι τέλη τα οποία θα είναι εύκολο να βαστάξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν έχετε άλλο χρόνο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχετε δίκιο ότι έχουμε λάβει μεγάλο αριθμό ισχυρισμών υγείας 4.600 από το 2008 που πρέπει να αξιολογηθούν. Ήδη τρεις παρτίδες τις έχουμε διεκπαιρεώσει και θα οριστικοποιήσουμε τις εργασίες μας εκτός από τα βοτανολογικά που μας ζήτησε η Επιτροπή μέχρι τέλος Ιουνίου ούτως ώστε η Επιτροπή να μπορέσει να κάνει μια πρόταση με βάση τη δική μας επιστημονική γνώμη. Ήθελα να πω όμως ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με παρτίδες, με δέσμες ισχυρισμών για τους ισχυρισμούς υγείας. Συνεχίζουμε ε, και βάσει του άρθρου 13.1 και βάσει του συστήματος αιτήσεων. Φέτος, παραδείγματος χάρη, λάβαμε 400 αιτήσει ε, βάσει του 13.5 και του 13.2 και αυτό αντιπροσωπεύει σημαντικό όγκο εργασίας, άρα ίσως να χρειαστεί επιβολή τελών. Και όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή, έχετε δίκιο, όταν θα έχουμε ε, αυτή την εφαρμογή, θα δούμε κατά πόσο μπορεί να γίνει και μια μελέτη αξιολόγηση για την επιβολή τελών από την ΕΦΣΑ. Συμπληρωματική ερώτηση για την αξιολόγηση αυτή Χρειάζεται φαντάζομαι ε, και επιπλέον προσωπικό γιατί όταν μιλάτε για 4.600 ε, ισχυρισμούς υγείας και νέους ισχυρισμούς που προέρχουν θα μειωθεί το προσωπικό, θα παραμείνει το προσωπικό το οποίο ασχολήθηκε με αυτά τα θέματα γιατί θα ασχοληθεί και στο μέλλον με κάτι παρόμοιο. Τι θα κάνετε. Όταν ήρθα στον Οργανισμό για την Ασφάλεια των Τροφίμων, μου είπαν ότι ήμουν άτυχη για το 2007 και μετά το 2008 και 2009. Θα ήταν τα δύο χρόνια κατά τα οποία θα είχαμε έργο εχμής, μεγάλο φόρτο εργασίας από την ΕΦΣΕ και ομολογώ ότι κάθε χρόνο αυξάνεται η εργασία μας. Δεν νομίζω λοιπόν ότι όταν ολοκληρώσουμε τις εργασίες για τον κατάλογο του άρθρου 13.1 θα έχουμε ολοκληρώσει το έργο μας για τους ισχυρισμούς γενικότερα και για άλλα θέματα που έχουν σχέση με τη διατροφή. Όπως σας είπα, συνεχίσουμε να λαμβάνουμε και νέες αιτήσει για τους ισχυρισμούς και γνωρίζουμε ότι στο άρθρο 13.1, στον κατάλογο αυτό, κάποιοι φορείς, κάποια, κάποιες μπορεί να επανέλθουν και να επανυποβάλλουν ισχυρισμούς για τις οποίους μπορεί να έχουμε δώσει αρνητική γνώμη ή αμφιλεγόμενη γνώμη και επίσης για τα θέματα διεκτικού κινδύνου είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τις ευρωπαϊκές ε, πολιτικές. Επομένως πρέπει εμείς να διατηρήσουμε τη δυνατότητά μας να δίνουμε επιστημονικές συμβουλές για να υποστηρίζουμε το έργο αυτών οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις. Ευχαριστώ. Ο κ. Αρσένης. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση για τα θέματα ισοδυναμίας. Είναι μια ερώτηση η οποία έχει τεθεί και για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, αλλά είναι ε, κάτι το οποίο αμφισβητείται από την επιστημονική κοινότητα, δηλαδή ότι οι γενετικά ε, ε, τροποποιημένοι οργανισμοί είναι ισοδύναμοι με άλλους συμβατικούς οργανισμούς, αν θέλετε. Όμως, υπάρχει, είναι διαφορετική ποιότητα, είναι, έχουν άλλη περιεκτικότητα σε βιταμίνες κτλ. Τι προτίθεστε να κάνετε με το θέμα αυτό. Θα αντικαταστήσατε την αρχή αυτή με τι. Ευχαριστώ. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι αναπτύχθηκε μια συγκεκριμένη ε, μεθοδολογία αξιολόγηση των κινδύνων για τους γενετικά μηχανισμένους οργανισμούς. Δεν μπορείς να αξιολογήσεις ε, ένα φυτό με τον ίδιο τρόπο που αξιολογείς ένα χημικό συστατικό. Και το ίδιο συμβαίνει και όταν συγκρίνει ένα γενετικά ένα φυτό με ένα συμβατικό φυτό. Στην ΕΦΣΑ και εγώ συνειδητοποιούμε ότι πολλοί τη χρησιμοποιούν αυτή τη μεθοδολογία, έστω και αν δεν την ε, ε, επικυρώνουμε. Όμως γίνεται μια επιστημονική συζήτηση με αυτούς που αμφισβητούν τη μεθοδολογία αυτή. Γι' αυτό το 2011 θέλω εφόσον ολοκληρώσουμε το έγγραφο, το κατευθυντήριο για, το, για τις τροφές και τις ζωοτροφές, μια και αλλάζουμε το κομμάτι που αφορά τα συγκριτικά στατικά, θέλουμε να οργανώσουμε ένα επιστημονικό εργαστήρι όπου θα ε, προσκαλέσουμε επιστήμονες από τα κράτη-μέλη, από με κυβερνητικούς οργανισμούς ε, και να κάνουμε μια αξιολόγηση αυτής της σύγκρισης αν θέλετε. Έτσι ώστε η συζήτηση η οποία γίνεται στην κοινή γνώμη και στην κοινωνία γενικότερα να αποτελέσει μια ευκαιρία για να το συζητήσουμε το θέμα με επιστήμονες που προέρχονται από όλους τους τομείς. Και αφού το συζητήσουμε θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Μια άλλη ερώτηση. Λαμβάνοντας υπόψη την κριτική που ασκήθηκε για, την, για τον ανεξαρτησία του προσωπικού της ΕΦΣΑ, ε, μπορείτε να επιβεβαιώσετε τι θητεία στην Εύσα, δεν θα ανδεχτείτε ε, άμεσα ή έμεσα κάποια θέση που να ασχολείται με την ε, βιομηχανία, την βιοτεχνολογία. Ναι, ναι, ε, εννοείται εγώ προσωπικά. Όχι, όχι. Δεν προτίθεμαι να απασχοληθώ από κάποια επιχείρηση τέτοια, από κάποια εταιρεία. Θα πρέπει να ξέρετε ότι στην ΕΦΣΑ έχουμε ένα καταστατικό, το οποίο εφαρμόζουμε και μας δεσμεύει όπως και όλοι οι υπάλληλοι των, των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει τα επόμενα, αφού φύγουμε από την ΕΦΣΑ να ε, ενημερώνουμε για το τι θα κάνουμε και πού θα πάμε και να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων. Προσωπικά όμως δεν νομίζω ότι θα μπω κάποια τέτοια, θα προσληφθώ από κάποια επιχείρηση ε, αν θέλετε μορφής. Δεν ενδιαφέρονται και για τις ε, και για τις ικανότητές μου. Η Φρανσουάς Γκροστέτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ συζητήσαμε πολύ για την αύξηση εργασίας, για τα προβλήματα, για τα ερωτήματα, σύγκρουση συμφερόντων, διαφάνειας κτλ. Μήπως θα έπρεπε τότε αντί να έχουμε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες να έχουμε εσωτερικούς εμπειρογνώμονες. Βέβαια δεν είναι έγκαιρη η ερώτηση γιατί θα πρέπει να αυξήσουμε τον προπολογισμό και τα κονδύλια για την υγεία δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα. Ε, έχετε κάνει όμως μια αξιολόγηση όσον αφορά τους δημοσιονομικούς και τους ανθρώπινους πόρους για αυτό το θέμα. Και δεύτερη ερώτηση που η κυρία Σουλή θα ήθελε να θέσει για, την, ε, ε, για το εμπόριο των, τροφίμων που, που τέθηκε το θέμα αυτό στον, τον Οκτώβριο. υπάρχουν, υπάρχει τόσο, μεγάλη ποσότητα ε, τροφίμων που είναι ακατάλληλα για βρώση και που κυκλοφορούν στο εμπόριο, μήπως θα πρέπει η ΕΕ να κάνει κάποια βήματα έτσι ώστε και οι κυβερνητικές, οργαν... και οι κυβερνητικές υπηρεσίες των κρατών μελών να καταπολεμήσουν το εμπόριο αυτό. Για το πρώτο σας ερώτημα πιστεύω ότι αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Δηλαδή ότι όντως θα πρέπει να διευρύνουμε την, ε, τις δυνατότητές μας για εσωτερική ε, αξιολόγηση αν θέλετε και να έχουμε εσωτερικούς εμπειρογνώμονες και προσπαθούμε να διευρύνουμε τον ε, προϋπολογισμό μας. Βέβαια, η ασφάλεια τροφίμων είναι ένα θέμα πολύ ψηλά στην στις προτεραιότητές μας, γι' αυτό θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την δημόσια υγεία θεωρούμε ότι αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις όσον αφορά τις, ε, τον αυξανόμενο αριθμό των αιτήσεων, θα πρέπει να διπλασιάσουμε τον αριθμό ε, του προσωπικού που ασχολείται με αυτές τις δραστηριότητε στην ΕΦΣΑ, που είναι περίπου 120-150 άτομα. Ξέρω ότι σας φαίνονται μεγάλος αριθμός, αλλά εάν συγκριθούμε με άλλες υπηρεσίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, που, ότι διαχειριζόμαστε στο τεράστιο αριθμό αιτήσεων, όπως πρέπει χάρη για, την, για τα φάρμακα, δεν είναι μεγάλο το προσωπικό. Ο αγροδιατροφικός τομέας είναι ο πρώτος οικονομικός τομέας στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε και η διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντική για την υγεία μας και για τη ζωή μας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τα επόμενα πέντε χρόνια να ε, διευρύνουμε τον προπολογισμό Τη ΕΦΣΑ κατά 50 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι τεράστιο ποσό εάν το συγκρίνουμε με τον τεράστιο αριθμό συμβουλών που, ε, που ε, επεξεργαζόμαστε και λαμβάνοντας υπόψη και, την, ε, και, τις καινοτομίες και το τις καινοτομίες που μας απασχολεί. Τώρα όσον αφορά την διακίνηση τροφίμων, ακατάλληλων τροφίμων, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συνδέεται περισσότερο με την ε, διαχείριση των κινδύνων και με τις αρχές που αφορά τις αρχές συμμόρφωσης, τις αρμόδιες αρχές συμμόρφωσης. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε εμείς είναι ότι αν μας το ζητήσουν μπορούμε να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε να εντοπίσουμε ε, τους αναδιόμενους κινδύνους, τα αναδιόμενα θέματα. Γι' αυτό έχουμε συστήσει μια μικρή ομάδα όπου ασχολούμεθα ε, με προϊόντα τα οποία δεν ε, αποτελούν αντικείμενο πολλής λεπτομερούς ρύθμισης, διότι πρέπει να ξέρουμε ότι τα τρόφιμα και ό,τι, ό,τι εμπορεύεται είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ένωση, διότι είμαστε μεγάλος εμπορικός εταίρος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το πρώτο ερώτημα μας είπατε ότι θέλετε να αυξηθεί ο προπολογισμό κατά 50 εκατομμύρια, λέει η κυρία Γκροστέτα, για να μπορέσετε να λειτουργήσετε κάτω από κανονικές συνθήκες. Εάν δεν σας δώσουν αυτή την αύξηση, γιατί ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι λίγο σφιχτά. Ε, εντάξει, μπορούμε να ελπίζουμε για τα επόμενα χρόνια, αλλά σήμερα είναι δύσκολο. Πιστεύετε ότι μπορείτε να ασκήσετε και να φέρετε εις πέρα στην αποστολή σας σωστά με τα χρήματα που έχετε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή σας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, γιατί είναι λίγο απεσιόδοξη η προσέγγιση. Αλλά ας προσπαθήσουμε. Θα πρέπει να δούμε τι βλέπουμε σαν προτεραιότητα εδώ. Ή μπορούμε να πούμε ότι το πιο σημαντικό είναι να ε, υποβάλουμε τις απαντήσεις μας εν στις διάφορες αιτήσει, χωρίς να, κάνουμε, να μπούμε στον κόπο να κάνουμε κάποιο διάλογο με τους ετούντες. Και μετά να συνεχίσουμε, ή να, να μετα, μεταφέρουμε κονδύλια από τις, ε, από τις ε, ασθένειες των ζώων, από, τους, από τις ουσίες που μολύνουν κτλ. σε άλλα θέματα. Γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ποια είναι τα σημαντικά θέματα για τα χημικά ας πούμε. Ή μπορούμε να πούμε όχι, θα πρέπει εμείς να ασχολούμεθα με τους πιο σημαντικούς τομείς και θα κάνουμε τη δουλειά μας, διότι αυτό που μας ε, ε, απασχολεί είναι η δημόσια ασφάλεια και η υγεία. Ασφάλεια τροφίμων και η δημόσια υγεία. και θα έχουμε μια περιορισμένη διαβούλευση, αν θέλετε, και αλληλεπίδραση με τους ετούντες. Yes, thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, we've heard a lot in this... Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντελάγκε. Ακούσαμε πολλά για τους ε, οικονομικούς πόρους και για τους πόρους γενικότερα και άκουσα πολύ τα απειλητικά που ακούμε ότι αν δεν έχουμε το προσωπικό και δεν έχουμε τους πόρους δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους καταναλωτές στην Ευρώπη. Αυτό που δεν άκουσα όμως είναι κάτι που αφορά το βασικό ερώτημα του πώς μπορεί να γίνει ΕΦΣΑ πιο αποτελεσματική βελτιώνοντας τις διαδικασίες οι οποίες δεν θα απαιτούν αναγκαστικά τόσο περισσότερους οικονομικούς πόρους. Παραδείγματος χάρη στον τομέα της βελτίωσης της επικοινωνίας και της συνεργασίας με τους ετούντες για την περίπτωση των ισχυρισμών υγείας. Οι διαδικασίες είναι και και χρονοβόρες και δαπανηρές και στο τέλος παίρνουν ένα ναι, ένα όχι. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να σηκώσει κανείς το τηλέφωνο και να πει έχω εδώ το φάκελό σας, είναι 95% τέλειος αλλά μας λείπει η πληροφορία για αυτό, για εκείνο και για τα άλλο. Μπορείτε να μας δώσετε αυτές τις πληροφορίες αντί να καταλήξετε σε ένα ναι ή ένα όχι και αν είναι όχι αυτοί οι άνθρωποι θα χρειαστεί να ξαναμπούν ξανά στην ακριβή διαδικασία και, που είναι και χρονοβόρο για εσάς. Πώς μπορείτε να βελτιώσετε λοιπόν τις διαδικασίες. Είναι σημαντικό να δούμε ότι δεν λέμε απλώς ναι ή όχι και έχουμε αλληλεπίδραση με τους ετούντες, αλλά περιορίζουμε τις επαφές μας, ε, διότι έχουμε τεράστιο αριθμό ισχυρισμών, ένα τεράστιο αριθμό αιτήσεων. Βεβαίως η επικοινωνία με τους ετούντες επηρεάζεται από την ε, έλλειψη πόρων και παράλληλα πρέπει να πούμε ότι δεν ε, ζητάμε υποστήριξη χωρίς να υποστηρίζουμε εμείς οι ίδιοι αυτά τα οποία κάνουμε και έχουμε σημαντικά προγράμματα με την υποστήριξη ενός εξωτερικού συμβούλου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας μας ε, και για να γίνουν πιο δυναμικές οι διαδικασίες μας ε, και να γίνουμε συνολικά περισσότερο αποδοτικοί και να χρησιμοποιήσουμε κατά το βέλτιστο τρόπο τους πόρους μας. Δεν θέλω να δημιουργήσω κανένα περιττό φόβο για τους πόρους που ζητάμε ή που δεν έχουμε, Απλώς ε, είπα ότι δεν μας υποστηρίζουν εξίσου με άλλους φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χειρίζονται παρόμοιο αριθμό αιτήσεων. 800 αιτήσει κάθε χρόνο είναι πολλέ και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε αυτό το φόρτο εργασία και να κρίνουμε το πού θα αποδώσουμε πόρου ανάλογα με το πού τοποθετούμε προτεραιότητε. Πάντω η ΕΦΣΑ θα είναι στην υπηρεσία σα και θα σα δώσουμε αυτά τα οποία μα ζητάτε, αλλά είναι σημαντικό να γίνεται αυτή η ανοιχτή συζήτηση. Λέμε ότι θέλουμε να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, ιδίω σε σχέση με του ετούντε, αλλά αυτό σαφώ έχει επίπτωση και επί των πόρων μα συμπληρωματική ερώτηση. Είναι η παλιά ερώτηση του αν το αυγό έκανε την κότα ή κότα το αυγό. Θα ξανακάνω την ερώτηση. Δεδομένου ότι υπάρχει αυτό ο ρυθμό των αιτήσεων, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να αυξηθεί ο προπολογισμό στην τρέχουσα περίοδο, εσεί γνωρίζετε τι διαδικασίε σα καλύτερα. Πείτε μα λοιπόν πού ακριβώ ε, ήταν η ερώτησή μου, μπορείτε να κάνετε αλλαγέ στι διαδικασίε σα και αν είστε πρόθυμοι να αλλάξετε τι διαδικασίε σα. Ναι, είμαστε πρόθυμοι να αλλάξουμε τις διαδικασίες μας. Είμαστε πρόθυμοι και έχουμε ήδη κάνει πολλές προσπάθειες. Το 2011 ε, θα εμφανίζεται καλύτερα και στο οργανόγραμμά μας το πώς αξιολογούμε και επεξεργαζόμαστε τις αιτήσει και εδώ έχουμε μια ομάδα, μια task force που θα χρησιμοποιείται ως ομάδα που θα μας βοηθά στον καλύτερο διάλογο με τους ετούντες. Αυτό θα είναι ένα πρώτο πρακτικό βήμα. Επίσης, χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο το μηχανισμό ε, μηδενισμού του χρόνου που είναι διαθέσιμος για να δίνουμε συγκεκριμένο χρόνο στους ετούντες. Επομένως βελτιώνουμε τις διαδικασίες μας και είμαστε πρόθυμοι να τις βελτιώσουμε κι άλλο και θα το κάνουμε και το 2011. Ευχαριστώ κυρία Γκουτιέρης Κορτίνας. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ κυρία Ζεσλέ Λανέλ. Μ' αρέσει ο τρόπος που απαντάτε και που βασίζετε τις απαντήσεις σας στην επιστήμη και δεν παρασύρεστε από το συνέστημα. Πρώτον, στην Ισπανία μας ανησυχεί πάρα πολύ η εισαγωγή προϊόντων που μας έρχονται από το Μαρόκο και που δεν υποβάλλονται προηγουμένως σε έλεγχο για να δούμε τι εντομοκτώνε, τι σπόροι χρησιμοποιούνται γι' αυτά. Όταν λοιπόν ελέγχει τις ποσοστώσεις η Ευρώπη, ξέρουμε ότι υπάρχει μια ποσότητα που δεν ελέγχεται. Η ΕΦΣΑ τι μπορεί να κάνει για την ανάλυση των προϊόντων αυτών που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Προϊόντα που μας έρχονται από το Μαρόκο και μπαίνουν στην ε, δικιά μας ε, αγορά τροφίμων. Δεύτερον, έχετε πληροφορίες για το ότι τι βαθμό συνδέονται οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί με τα οντομοκτώνα. So on the first question, which Για το πρώτο, για τις εισαγωγές. Εμείς ε, δεν ευθυνόμαστε για τον έλεγχο των εισαγωγών, όμως συνηθίζεται τελευταία η Επιτροπή να μας ζητάει επιστημονική αρρωγή κάθε φορά που πρόκειται για ένα προϊόν που μπαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά και όπου εντοπίζεται ένα χημικός παράγοντας που μολύνει τα τρόφιμα, υπάρχει υποψία για κάτι τέτοιο. Και όντω από το 2007 συνεισφέρουμε κι εμείς σε αυτό και έτσι έχουμε αναπτύξει κάποιες διαδικασίες οι οποίες μας επιτρέπουν μέσα σε λίγε μέρες να δώσουμε μία επιστημονική γνωμοδότηση για να βοηθήσουμε την αξιολόγηση κινδύνου όταν υπάρχει κάποιο κίνδυνο για τη μελαμίνη, για παράδειγμα, για την νοικοτήνη, επίση τα μανιτάρια που μα έρχονται από την Κίνα ή ακόμα και στο χείριο κρέα από την ε, Ιρλανδία με τοξίνε. Και γενικά προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να αποφύγουμε κρίσεις για τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς. Δεν μπορούμε να δώσουμε έτσι γενικά μια απάντηση. Πρέπει να δούμε εξειδικευμένα για τον κάθε γενετικά τροποποιημένο οργανισμό. Όντως, κάποιοι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί ε, φτιάχνονται για να περιοριστεί η χρήση εντομοκτώνων ακριβώς. Στα πλαίσια της υπάρχουσας νομοθεσίας στην Ευρώπη είναι πληροφορία που παίρνουμε στους φακέλους μας, αλλά δεν είναι αρμοδιότητά μας να αξιολογούμε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για τα αποτελέσματα ή για τα ωφέλη στο περιβάλλον από γενετικά τροπομένους οργανισμούς. Στο μέλλον μπορεί. Προς το παρόν δεν είναι αποστολή μας. Για κάποια προσθετικά, ναι. Για τα ντομοκτώνα, ναι, είναι αρμοδιότητά μας. Αλλά δεν μας έχει δοθεί τέτοια ευθύνη όσον αφορά τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ευχαριστώ. Συγκροματική ερώτηση. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μου απαντήσετε. Δηλαδή, δεν έχετε ευθύνη για τα εισαγόμενα προϊόντα δεδομένου του όγκου των προϊόντων που μας ε, έρχονται και από άλλες χώρες της Μεσογείου στα πλαίσια των συμφωνιών ε, εμπορίας που έχουμε με άλλες χώρες. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποια υπηρεσία που ελέγχει τα προϊόντα αυτά όλο και περισσότερο, όλο και πιο μαζικά θα μας έρχονται από τη Βόρεια Αφρική εδώ στην Ευρώπη. Απάντηση. Ναι. Ήδη στον τομέα τροφίμων, όπως και σε ένα, άλλο, σε ένα σωρό άλλους τομείς, έχουμε την παγκοσμιοποίηση. Και πρέπει να σας πω ότι το σύστημα, το Ευρωπαϊκό Ασφάλειας Τροφίμων, προσπαθεί να θέσει εφαρμογή μηχανισμούς, ρυθμίσεις, αλλά και σώματα, υπηρεσίες που να είναι αρμόδιες για τα προϊόντα αυτά, ώστε να μην έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών μας. Ως εύσα πάντως, εδώ πρέπει να σας απαντήσω ότι έχουμε εκπονήσει ένα σύστημα με μια μικρή ομάδα όπου προσπαθούμε να ελέγξουμε τι γίνεται με τα μη ρυθμισμένα προϊόντα. Έτσι, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι έγκαιρα μπορούμε να εντοπίσουμε δυνητικούς κινδύνους. Και αν κάτι συμβεί, το σημαντικό είναι ότι είμαστε στην υπηρεσία σας και της Κομισιόν γρήγορα να γνωμοδοτήσουμε ώστε να ληφθούν μέτρα και να προστατευτούν οι καταναλωτές. Ευχαριστούμε. Να σας Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ξέρετε υπάρχουν δύο επιδημίες Παχυσαρκία και διαβήτη που είναι πάρα πολύ ε, σημαντικές και οφείλω να μιλήσω ότι επηρεάζουν ιδιαίτερα ε, γιατί είναι το μέλλον αν θέλετε της, ε, του, πλανήτη μας. Η ΕΦΣΑ προωθεί το θέμα της υγιεινής διατροφής. Ξέρω ότι τα πράγματα είναι δύσκολο, αλλά θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι ένα τομέα τη αρμοδιότητά σα. Αλλά λόγω των, ε, του προπολογισμού και τα λοιπά, τι πρεσβεύεται. Ναι, όντω ε, η διατροφή είναι ανήκει στους, αρμοδιότητε μα. μας, ε, έχουμε ένα ρόλο σύμφωνα με τι εντολές που μα έχει δοθεί και πρέπει να δίνουμε συμβουλές για να βοηθήσουμε και αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο να έχουν ε, τις σωστές ε, πληροφορίες στη διάθεσή τους. Έχουμε εξετάσει τα χαρακτηριστικά πολλών ε, διατροφικών συστατικών. Θα έχουμε βοηθήσει τις, τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν μια σωστή μεθοδολογία για να μετατρέψουν ε, την, ε, τα συστατικά σε σωστή διατροφή, διότι δεν τρώμε συστατικά, ε, τρώμε τρόφιμα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ο ρόλος μας είναι να βοηθήσουμε στον τομέα αυτό περαιτέρω. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν συμπληρωματικές ερωτήσεις. Κύριο Σταταρέλε, Όπως είδατε κυρία μου από τις διάφορες ερωτήσεις που ετέθησαν, η Επιτροπή αυτή εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή τα, της εργασίας ΕΦΣΑ. Και σήμερα το πρωί στην έκθεση Μπερλάτο εγκρίναμε μια τροπολογία που θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της ΕΦΣΑ στην, στην κοινοποίηση των κινδύνων που αφορούν τη διατροφική αλυσίδα και εκφράσαμε την επιθυμία όλα τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν αντίστοιχους εθνικούς οργανισμούς με σκοπό τη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Στην Ιταλία παρά την ύπαρξη ενός προηγουμένου νόμου που προέβλεπε την δημιουργία ενός εθνικού οργανισμού, ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί αυτός ο οργανισμός. Εγώ προφανώς δεν σας ζητάω την ε, γνώμη σας για την νομοθεσία ενός κράτους μέλους, δεν ανήκει αυτό στις αρμοδιότητές σας, αλλά μία τεχνική αξιολόγηση θα ήθελα να κάνετε, μια και είστε ένα τρίτο άτομο αν θέλετε εσείς. Με βάση την ερμηνεία, την εμπειρία σας, ε, η δημιουργία ενός εθνικού οργανισμού ε, που θα συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό θα μπορούσε να βοηθήσει στην οργάνωση των εργασιών σας. Ευχαριστώ. Είναι σαφές ότι υπάρχουν τελείως διαφορετικά συστήματα στα κράτη-μέλη και κάποια από αυτά, 10-12, έχουν ε, εθνικούς οργανισμούς για την διατροφική ασφάλεια και άλλα όργανα αξιολόγησης των κινδύνου. Άλλα κράτη-μέλη δεν, έχει, δεν έχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνεργαζόμαστε με έναν αποτελεσματικό τρόπο. Και ε, μια και μιλάτε για την Ιταλία, να σας πω ότι έχουμε μια πολύ αποτελεσματική συνεργασία με την Ιταλία. Είναι ένα από τα κράτη-μέλη που ε, είναι τα πιο δραστήρια όσον αφορά τον ε, αριθμό των χορηγιών των ε, που έχουμε όσον αφορά την αξιολόγηση των κινδύνων. Φαίνεται επομένως ότι δεν υπάρχει ένα θεσμικό μοντέλο. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι η θέληση. Η θέληση, η πραγματική θέληση του κράτους μέλους να συνεργαστεί μαζί μας έτσι ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη, να υπάρχει συνεργασία έτσι ώστε να βελτιώσουμε τη δημόσια υγεία. Okay. Ωραία, περνάμε στον τρίτο γύρο ερωτήσεων. Δεν έχουμε μία εγγεγραμμένο μέλο, δεν έχουμε δεύτερο άτομο από την ομάδα ECR. Επόμενη ερώτηση από του Πρασίνου, Καρλ Σούιτερ. Ευχαριστώ πολύ συζητήσαμε τα θέματα των εμπειρογνωμόνων πρέπει να είναι ανεξάρτητοι κλπ. Και η αξιολόγηση κινδύνου είναι θέμα στο οποίο έχει ασκηθεί κριτική και στο παρελθόν. Πίσω σας κάθομαι για να με δείτε. Λοιπόν, ε, για το τελευταίο αεραβόσιτο που είχατε την ευκαιρία να δώσετε επιστημονική γνωμοδότηση που βασίζεται ε, σε συνδυασμό προηγουμένων γενετικώς τροποποιημένων φυτών και σε ολόκληρη τη μελέτη λέγεται ότι δεν είναι πιθανόν ότι θα αλλάξει το κατά πόσο είναι αλλεργιογόνο, δεν είναι πιθανόν ότι θα αλλάξει η τοξικότητα, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι όταν φτάνουμε στην ε, τοξικότητα, η προσθήκη πολλών ουσιών μπορεί να μην μας κάνει απλώς το άθροισμά τους, το ενα συν 1 συν 1 συν 1, να μην κάνει απλώς τέσσερα δηλαδή. Και ε, σε σχέση με τη μελέτη αυτή, εκτός από τη ε, μελέτη σε νεοσούς 42 ημερών για τις ζωοτροφές, είναι πολύ μικρός ο χρόνος κατά τον οποίο τρέφονται ε, η νέωση οι 42 ημέρες. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την αξιολόγηση κινδύνου την οποία κάνετε. Πώς μπορείτε να είστε ικανοποιημένοι από αυτά τα οποία έχετε κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν ε, για τις αβεβαιότητες ε, και για το ότι πολλές φορές, όπως είπατε, χρησιμοποιούμε τη λέξη unlikely, ότι δεν είναι πιθανόν ότι θα γίνει κάτι. Αυτό το οποίο λέμε είναι αυτό το οποίο μπορούμε να πάρουμε από την κατάσταση των πραγμάτων, από την επιστήμη και από την επιστημονική γνώση που έχουμε. Τούτου λεχθέντος, οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν κάνουμε αξιολόγηση κινδύνου πριν από τη θέση σε εμπορία του προϊόντος, αλλά επίσης δίνουμε τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθείται ο κίνδυνος, ούτως ώστε κάποια επίπτωση που δεν ε, ήταν αρχικά αναμενόμενη ε, μπορεί να εξεταστεί κατά, την, ε, κατά το σύστημα αξιολόγησης post-mortem, όπως το αποκαλούμε. Είναι κάτι το οποίο βασίζουμε και σε αιτήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητάει η Επιτροπή κάθε χρόνο η ΕΦΣΑ να δίνει μια επιστημονική έκθεση όπου αξιολογούμε τα δεδομένα που λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη και από τις εταιρείες ε, γενετικά τροποποιημένων προϊόντων σε σχέση με αυτά τα οποία παρατηρήθηκαν στην πράξη για να δούμε αν υπάρχει κάποια επίπτωση που δεν ήταν αρχικά αναμενόμενη ή αν η δυνητική κίνδυνη που είχαμε εντοπίσει όντως ε, στην πράξη αποκαλύφθηκε ότι υλοποιήθηκαν. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη μου απάντηση. Για τις ε, δοκιμές ε, από τη χορήγηση ζωοτροφών σε νεοσούς δεν έχουμε αποκλείσει τέτοιου είδους δοκιμές. Έχουμε πει ότι μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις όταν συγκρίνουμε ισοδύναμα μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και περαιτέρω τοξικολογικές μελέτες και ακριβώς αυτό θέλουμε να συζητήσουμε σε αυτό το σεμινάριο το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως και ελπίζω ότι θα έχουμε ενεργό συμμετοχή από εμπειρογνώμονες για να συζητήσουμε το θέμα αυτό το Μάρτιο του 2011. Και για τις αξιολογήσεις κινδύνου για το περιβάλλον προσφάτως ε, ε, ε, με βάση αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάναμε μια αναθεώρηση για να προσαρμόσουμε την μεθοδολογία μας και να αξιολογήσουμε το τη μακροπρόθεσμη επίπτωση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών επί του περιβάλλοντος. Αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να συγκεντρώσουμε περισσότερα δεδομένα και να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε και τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον στον τομέα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση του κ. Σλίτερ. Δέκα δευτερόλεπτα μόνο. Καταλαβαίνω ότι εμείς είμαστε τα ειδικά χειρίδια. Γιατί δεν ζητάτε μια ε, νέα δοκιμή όταν είναι κάτι καινούριο. Και όταν υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές τοξίνες σε ένα φυτό, γιατί δεν ζητάτε και συμπληρωματικούς ελέγχους. Γιατί η αρχική χορήγηση στροφών για τον έλεγχο ήταν πολύ βραχυπρόθεσμη και έγινε μόνο για να ελεγχθούν οι διατροφικές ιδιότητες. Απάντηση. Νομίζω ότι δεν αντανακλά την πραγματικότητα το να πούμε ότι δεν ε, χρησιμοποιούμε τη δυνατότητα του να κάνουμε δοκιμές 90 ημερών, γιατί και αυτό έχει γίνει. Αυτό που είπα είναι ότι Πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται από την αρχή να ζητάμε τέτοιες δοκιμές χορήγησης ζωοτροφών συστηματικά και χρησιμοποιήσαμε το κριτήριο του πότε καθίσταται σημαντική μια τέτοια δοκίμη. Πάντως είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση, έχουμε πολλούς εμπειρογνώμονες από πολλές διαφορετικές προελεύσεις για αυτό το θέμα και θα το συζητήσουμε το 2011 στο σεμινάριο που ανέφερα. Φρεντερικ Ρίς. Ευχαριστώ. Τουλάχιστον 10 ερωτήσει τέθηκαν για το θέμα τη ανεξαρτησία ε, των επιστημονικών εμπειρογνωμόνων, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι και ένα από του κύριου λόγου ύπαρξή μα το να σα κάνουμε τέτοιε ερωτήσει. Αντί λοιπόν για άλλη μια φορά να μιλήσουμε για τι αρχέ, σα δούμε μια περίπτωση. Μπισφενόλ Α που δεν αναφέρθηκε και καλύτερα γιατί είναι δύσκολο όταν κανείς παίρνει το λόγο τόσο αργά στη συζήτηση. Η Επιτροπή θα το απαγορεύσει, η πρόταση θα γίνει το Μάρτιο νομίζω ή Φεβρουάριο βάσει γνωμοδότησης από την δικιά σας την υπηρεσία που είναι έτσι κάπως χλιαρή. Τώρα, Μπορεί να επανέλθετε βέβαια σε αυτό το θέμα. Εμείς οργανώνουμε ακρόαση, με, μάλλον οργανώσαμε την Κορίν Πάζια ε, μια ακρόαση και μόνο δύο είπαν ότι είναι αυλαβές για την παρουσία δηλαδή της ουσίας αυτής στα πιπερών. Ένα μέλος του πάνελ σας ήταν στη μειοψηφία. Εσείς πώς αναλύετε αυτό το θέμα του πιφενόλ που μας απασχόλησε και θα απασχολήσει και μας εδώ στις αρχές επόμενης χρονιάς. Απάντηση. Είναι αλήθεια ότι το αρμόδιο πάνελ ασχολήθηκε έξι μήνες με αυτή την ουσία. Πολύ δηλαδή. Η επιστημονική μας γνωμοδότηση έλεγε ότι προηγουμένως είχαμε αναλύσει όλα όσα έχουν γραφτεί από επιστήμονες γι' αυτό και συγχρόνως λέμε ότι ότι δεν θα αναθεωρήσουμε την ημερήσια δόση. Όπως και άλλες υπηρεσίες και οργανισμοί στον κόσμο, διαπιστώσαμε κι εμείς ότι οι ορισμένες μελέτες μιλούν για επίπεδα, αλλά οι μελέτες αυτές έχουν και λήψεις. Εμείς τα αναφέραμε αυτά στην γνωμοδότησή μας. Και από εκεί και πέρα ο διαχειριστής κινδύνου παίρνει την απόφαση και εσείς είπατε ποια είναι η απόφαση αυτή. Είναι σημαντικό να πούμε εδώ ότι το εργαστήριο που οργανώθηκε από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πριν από μερικές εβδομάδες κατέληξε σε αντίστοιχα συμπεράσματα με τα δικά μας. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό για αυτό το θέμα είναι να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνουμε τις βεβαιότητές μας. Γιατί αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις πρέπει να ξέρουν σε τι βαθμό μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στην κατάσταση πραγμάτων έτσι όπως την περιγράφει η επιστήμη και να μπορούν να βασιστούν και στον κοινωνικό διάλογο που λαμβάνει η χώρα, ώστε να ξέρουν πού πρέπει να βάλουν περισσότερο βάρος. Και εδώ έρχεται και η αρχή της προφύλαξης. Έτσι λοιπόν εμείς στην ΕΦΣΑ Πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ελέγχουμε τις ερευνητικές εξελίξεις των επόμενων εβδομάδων και μηνών και να ξέρετε ότι εμείς έχουμε αναλύσει τη χημική ουσία που θα αντικαταστήσει την ουσία αυτή όταν θα απαγορευτεί στα μπιπερό. Γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι θα αντικατασταθεί από κάτι άλλο το οποίο είναι ασφαλές. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη θέση σας, αλλά βλέπετε εμείς θέλουμε στα πλαίσια της δικιά σας εντολής να διαπιστώνουμε ότι υπάρχει και κάποια τόλμη. Θυμάμαι στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος ε, συζητούσαμε για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και εκεί η συζήτηση πήγαινε προς κάθε κατεύθυνση. Τελικά η υπηρεσία όμως κατάφερε και προχώρησε. Αυτό περιμένουμε και από εσά. Συμπληρωματική ερώτηση όμως που έχει σχέση με αυτό. Αναφερθήκατε πολύ σύντομα στην αρχή όταν είπατε για το ευρωβαρόμετρο, ότι ο κόσμος και ε, θεσμικό όργανα και τα λοιπά σας ε, βλέπουν θετικά. Εγώ όμως δεν σας βλέπω πολύ παρόντες. Θα μου πείτε δεν είναι ο ρόλος σας να προβάλλεστε. Εγώ πιστεύω ότι ναι, γιατί εφόσον θέλετε να συμμετέχετε στις μεγάλες συζητήσεις που γίνονται στην κοινωνία, πώς θα επικεντρώσετε κάπως τις προσπάθειές σας και προς αυτή την κατεύθυνση. Απάντηση. Συμφωνώ μαζί σας για το ότι πρέπει με την επικοινωνία μας να είμαστε περισσότερο παρόντες. Και προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που επικοινωνούμε με τον κόσμο. Θα φροντίσουμε να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα ε, τους σπόρους μας και θα αναπτύξουμε μία πιο θεματική προσέγγιση στις, ε, στην επικοινωνία μας κυρίως εκεί που μπορούμε να εξηγήσουμε πώς επηρεάζει το έργο μας στη δημόσια υγεία. Θα εξηγήσουμε τι κάνουμε για τις ζωνώσεις, που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Στην Ευρώπη πιστεύω ότι έχουμε προχωρήσει πολύ στην μείωση των ζωνώσεων, της παρουσίας τους. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, για παράδειγμα, μπορούμε να εξηγήσουμε ποιο είναι ο ρόλος τη ΕΦΣΑ, τι έχει κάνει και πώς χρησιμοποιείται η γνωμοδότησή μας στο συγκεκριμένο θέμα από την επιστημονική κοινότητα, από τους διαχειριστές κινδύνου. Συνεπώς, δεν αλλάζει σημαντικά η επικοινωνία μας, αλλά ο τρόπος που επικοινωνούμε. Επίσης, το θέμα της ανεξαρτησίας θα είναι ένα θέμα σχετικά με το οποίο ε, πρέπει να επικοινωνήσουμε καλύτερα για να εξηγήσουμε γιατί βασιζόμαστε σε ανεξάρτητους επιστήμονες, γιατί πρέπει να υπάρχει η ανεξαρτησία αυτή και γιατί πρέπει να καταπολεμήσουμε κάθε σύγκρουση συμφερόντων. Και να εξηγήσουμε ότι δεν θέλουμε να συνεργαζόμαστε με επιστήμονες οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στη βιομηχανία. Είναι πράγματα που έχουν πάρει μεγάλη σημασία τον τελευταίο καιρό στην επιστημονική έρευνα. Λέντα Μακάβεν. Ευχαριστώ. Αποκαλείστε Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, αλλά το έργο σα καλύπτει και άλλου τομεί. Αναφέρετε περιβαλλοντικά θέματα και γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και κλωνοποίηση. Εξετάζετε θέματα για την ευζοία των ζώων. Η ισορροπία ποια είναι στο έργο σα. Θεωρείτε τον οργανισμό σα αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων. Καταρχήν, όταν κάνει σχόλια η Επιτροπή για την κλωνοποίηση, μα είπε η Επιτροπή ότι η ΕΦΣΑ είπε ότι είναι ασφαλέ, επομένω είναι ασφαλέ να το φάμε βλέπετε εσείς ε, να είναι ένα στοιχείο πιο σημαντικό από τα άλλα όταν παρουσιάζετε τις αποφάσεις για την κλωνοποίηση, για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, η ασφάλεια των τροφίμων, η περισχή του περιβάλλοντος ή της ε, υγιεινής των ζώων. Νομίζω ότι η ασφάλεια των τροφίμων και η επίπτωση της επί της ε, υγείας του ανθρώπου είναι η σημαντική αποστολή που μας έχει δοθεί και αυτό δικαιολογεί και τον τίτλο του φορέα μας. Όταν αξιολογούμε προϊόντα ή τεχνολογίες, ενδέχεται επιπροσθέτως να αξιολογήσουμε και κάτι άλλο. Και αυτό, όπως είπατε, έχει εξελιχθεί πολύ, γιατί έχουμε και την ευζοία των ζώων και το περιβάλλον, αποτελεσματικότητα κλπ. Αυτά όμως συμπεριλαμβάνονται σε μια συνεκτική τελική συμβουλή που ποτέ δεν λησμονεί ότι το σημαντικό μας έργο αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. Έτσι το βλέπουμε. Σχετικά με την ε, πολυτομεακή εμπειρογνωμοσύνη που έχουμε, που έχουμε βρει και από το προσωπικό μας και από τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, ε, πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να έχουμε αποτελέσματα και για την ασφάλεια των τροφίμων και για τα υπόλοιπα θέματα που εσείς ως διαχειριστές του κινδύνου, ως νομοθέτες, μας ζητάτε μια προσέγγιση γιατί εσείς χρειάζεστε να έχετε τη συνολική εικόνα. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε την ασφάλεια όταν εξετάζουμε την ευζοία των ζώων ή την αποτελεσματικότητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να συνεχίσουμε να το έχουμε στο επίκεντρο της εργασίας μας και στο μέλλον. Άρα ποτέ δεν εξετάζεται αν κάτι πρέπει να γίνει, το αν πρέπει να έχουμε κλωνοποιημένο κρέας, παραδείγματος χάρη και μετά από αυτό που είπε και η Julie Γκέρλινγκ ε, για τους εθνικούς φορείς ασφάλειας των τροφίμων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό που θα θέλαμε είναι να αντικαταστήσουμε τη δουλειά που γίνεται στα κράτη-μέλη. Γίνεται αυτό ή απλώς γίνεται επικάλυψη και διπλασιάζεται το κόστος μας αντί να εξοικονομούμε χρήματα με μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Δεν θα έλεγα ότι εξετάζουμε το επιθυμητό για ένα προϊόν ή για μια τεχνολογία, αλλά όταν παραδείγματος χάρη μας ζητούν να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα ενός προϊόντος, εξετάζουμε βέβαια το αν το προϊόν αυτό θα προσφέρει κάποιο όφελος είτε στους αγρότες που θα το χρησιμοποιήσουν, είτε στα ζώα που θα το καταναλώσουν, είτε στο περιβάλλον, είτε στον καταναλωτή που θα καταναλώσει αυτό το προϊόν. Αυτό είναι πολύ παρόμοιο με αυτό που εσείς αποκαλέσατε το επιθυμητό της διαδικασίας. Είναι η δραστηριότητά μας ε, η οποία καλύπτει αυτό τον τομέα. Η δική μας συντολή είναι διαφορετική από αυτή που έχουν οι εθνικοί φορείς ασφάλειας τροφίμων και δεν νομίζω ότι υπάρχει ανταγωνισμός εδώ, διότι η ΕΦΣΑ ποτέ δεν πρόκειται να εξετάσει θέματα που αφορούν μόνο τοπικό ή μόνο εθνικό επίπεδο. Προφανώς αυτό δεν αποτελεί έργο της ΕΦΣΑ. Πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά τα οποία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενδιαφέρουν. Για να το κάνουμε όμως αυτό χρειαζόμαστε στοιχεία από τους Εθνικούς Φορείς Ασφάλειας των Τροφίμων, χρειαζόμαστε εμπειρογνώμονες από τις Εθνικές Αρχές και χρειαζόμαστε και πρόσβαση στην εμπειρογνωμοσύνη τους. Και γι' αυτό έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα βάσει του οποίου η ΕΦΣΑ βασίζεται στο έργο των Εθνικών Φορέων Ασφάλειας των Τροφίμων και στο μέλλον θα συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε. Ελιζαμπέτα Γκαρντίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Διευθύντρια. Πάρα πολλά πράγματα έχουν ήδη ληχθεί και σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μας δώσατε. Θα ήθελα όμως να επανέλθω για λίγο στη συζήτηση που γίνεται για αυτά τα αυτές τις αιτήσει. Γιατί πραγματικά υπάρχει μια πορεία για αυτά τα αιτήματα υγείας, ε, για την υγεία που... Για αυτές τις, ε, ε, τα, που θεωρούν ορισμένα πράγματα τα οποία ίσως βοηθούν ή κάτι... Θα ήθελα να ξέρω όλες αυτά, όλα αυτά τα οποία λέγονται, τα εξετάζετε ή όχι. Και λαμβάνοντας υπόψη και τον όγκο των, της εργασίας σας, ο οποίος αυξάνει και λαμβάνοντας υπόψη και τον κανονισμό για την ενημέρωση των καταναλωτών, πέραν της αύξησης του προϋπολογισμού ή του προσωπικού σας έχετε να κάνετε κάποια πρόταση στην Επιτροπή για την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς σας. για αυτούς τους ισχυρισμούς ε, για, τα, για την υγεία ε, το κάνουμε όλα αυτά το, τις, αξιολογούμε τους ισχυρισμούς μέσα στα πλαίσια της, ε, των αρμοδιοτήτων που έχουμε και προφανώς πρέπει να είμαστε σίγουροι και αυτό το επιβεβαιώνουμε ότι αυτοί οι ισχυρισμοί στηρίζονται σε, κάποιες, σε κάποια επιστημονικά δεδομένα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια εργαζόμεθα. Όμως έχουμε δημιουργήσει ένα, έχουμε συντάξει ένα κείμενο το οποίο βοηθάει και τους ετούντες στην βιομηχανία, ποια είναι οι απαιτήσει, τι θα τους ζητήσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε την αξιολόγησή μας και τους λέμε πώς αξιολογήσουμε και τα δεδομένα τα οποία θα μας στείλουν. Πιστεύω ότι η ερώτησή σας επίσης σχετίζεται με, το, με τη βελτίωση του διαλόγου με τους ετούντες. Δηλαδή ε, αυτοί οι οποίοι υποβάλλουν μια αίτηση και η οποία έχει απορριφθεί σε ένα πρώτο γύρο, τι θα γίνει, μπορούν να επανέλθουν και πόσο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει μια σειρά workshops που ξεκινάνε και αυτή την εβδομάδα, όπου έχουμε καλέσει εμπειρογνώμονες από την βιομηχανία για να ε, δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα εξετάσουμε κάποιους συγκεκριμένους ισχυρισμούς ε, για να δούμε ποιες είναι, ποια είναι τα επιστημονικά δεδομένα και για την διατροφική αξία και να γίνει μια ε, ανταλλαγή απόψε ανάμεσα στους επιστήμονες και στην βιομηχανία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύουμε, και για την ποιότητα των αιτήσεων που θα πάρουμε στο μέλλον. Τώρα για τους ισχυρισμούς συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με την Κομισιό για να είμαστε σίγουροι ότι ε, αυτά τα οποία λέμε είναι σωστά και η Κομισιό μας έχει βοηθήσει για να ορίσουμε τις προτεραιότητες ας πούμε σε αυτή τη στιγμή έχουμε σταματήσει τη δουλειά για τα βοτανολογικά ε, προϊόντα, βοτανολογικά προϊόντα, στα οποία θα επανέλθουμε αργότερα και πιστεύουμε ότι αυτή η αλληλεπίδραση είναι πάρα πολύ σημαντική για να είμαστε σίγουροι ότι όλη αυτή η δουλειά που είναι τεράστια θα ε, γίνει με ανταποτελεσματικό και επικοδομικό τρόπο από την ΕΦΣΑ. Τελευταίος γύρος ερωτήσεων, σοσιαλδημοκράτες, ε, ο Γιώργενσεν δεν είναι εδώ, η κυρία Ντάκμα Ροτμπέρεντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να επανέλθω λίγο στη βασική γραμμή της ακρόασης αυτής. Από τη μια μεριά εξετάζουμε την ποιότητα των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων. Εδώ Συζητήσαμε επίση και για του γενετικού κάτροπημένου οργανισμού και την ανεξαρτησία των εμπειρογνωμών. Το ξέρετε το θέμα. Εγώ την ξέρω την απάντηση, αλλά ίσω δεν την ξέρουν οι συνάδελφοι ή να θέλουν να την ακούσουν. Επαναλαμβάνω λοιπόν. πώ είσαστε σίγουροι ότι έχετε την καλύτερη επιστημονική πραγματογνωμοσύνη. πώ είσαστε σίγουροι ότι έχετε στην πάρμα του καλύτερου επιστήμονε, του πιο αποτελεσματικού Και πώ είσαστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι ε, τρώνε κάτι υγιεινό. Με την εντολή που έχετε και με τους ε, κανονισμούς που έχετε, που δεν έχουμε αλλάξει, πόσο δύσκολο είναι για σας να διευρύνετε τις αρμοδιότητές σας και να λάβετε υπόψη όλα όσα ζητάει η κοινωνία. Όχι μόνο δηλαδή την επιστημονική πραγματογνωμοσύνη, αλλά να, για τα κλωνοποιημένα ζώα, αν πρέπει να τα τρώμε ή όχι, ή άλλα πράγματα που επιστημονικά οι πολίτες μας ε, νιώθουν ότι χρειάζονται. Φτάσαμε στο τέλος του γύρου των ερωτήσεων και η Ντάγμα σχεδόν έκανε τη σύνοψη που θα έκανα εγώ. Η Επιτροπή μας ε, σαφώς ενδιαφέρεται για τα ε, είδη διατροφής και είναι αντικείμενο των εργασιών μας και μας ενδιαφέρει ε, η αξιολόγηση κινδύνου για τα διάφορα προϊόντα και το θέμα της ανεξαρτησίας της ΕΦΣΑ, της ποιότητας των γνωμοδοτήσεων, ε, η δυνατότητα του να δουλεύουμε προληπτικά Όλα αυτά είναι βασικά ερωτήματα, κύριο, ε, από τα οποία στράφηκαν και όλες οι ερωτήσεις μας. Τώρα έχετε πέντε λεπτά χρόνο να απαντήσετε συνολικά, κλείνοντας αυτό τον κύκλο θεμάτων ε, και δίνοντάς μας τις απαντήσεις σας. Ευχαριστούμε. Um, Ευχαριστώ πολύ. Όπως λέτε, Τάκμαρ, είναι δύσκολο. Αλλά έχουμε συγκεκριμένη αποστολή, σημαντική αποστολή στην ΕΦΣΑ. Να προστατεύσουμε, να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τους καταναλωτές, το περιβάλλον και να φροντίσουμε και για την προστασία των ζώων. Είμαστε καλά εξοπλισμένοι, πιστεύω. Η ΕΦΣΑ δεν είναι όπως ήταν πριν από πέντε χρόνια. Χάρη στην δικιά σας στήριξη μεταξύ άλλων, κάναμε πολλές προσπάθειες κι εμείς για να βελτιώσουμε την μεθοδολογία μας. Έχουμε περισσότερους πόρους, ευρύτερες διαδικασίες. Έχουμε σε ένα μεγάλο βαθμό βελτιώσει τη συνεργασία μας την επιστημονική με τις χώρες μέλη από το 2007 και μετά. Έχουμε διαφοροποιήσει επίσης εντυπωσιακά το εύρος της πραγματογνωμοσύνης στην οποία έχουμε πρόσβαση. Συγχρόνως όμως αναγνωρίζουμε ότι οι προκλήσεις είναι όλο και μεγαλύτερες, όλο και περισσότερες αιτήσει δεχόμαστε. Σας είπα, 900 φέτος το 2010 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διπλασιάστηκαν δηλαδή σε σχέση με πέρυσι. Αυτό πρέπει να αναγνωριστεί. Και αυτό θέλω να σας μεταφέρω εδώ. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τα καλύτερα δυνατόν αποτελέσματα. Και θέλουμε επίσης να φροντίσουμε να κάνουμε τη βέλτιστη χρήση των πόρων μας. Και επανέρχομαι σε αυτό που λέγαμε και πριν. Εδώ δεν είμαι για να ζητήσω παραπάνω λεφτά από εσά. Όχι, πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας τη σημασία που έχουν τα τρόφιμα στην καθημερινή μας ζωή και στην υγεία μας. Πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη μας την σημασία που έχει ο τομέας ε, της γεωργίας και των τροφίμων για την ευρωπαϊκή οικονομία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας επίσης ότι πρέπει να ανταποκριθούμε στις δικές σας ανάγκες που είναι διαχείριση κινδύνου. Όχι μόνο για την ασφάλεια, αλλά και για το περιβάλλον, για την αποτελεσματικότητα, για τα ωφέλη πράγματα τα οποία συζητιώνται σήμερα στην κοινωνία. Θέλουμε να είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε να παίρνετε τις αποφάσεις σας βασισμένοι στην επιστημονική γνώση. Γι' αυτό σας ζητάμε παραπάνω στήριξη. Κάνουμε εμείς πάντως προσπάθειες για να ανταποκριθούμε στις δικές σας ανησυχίες βάσει των ερωτήσεων που θέσατε για τη διαφάνεια, για τον τρόπο που διατυπώνουμε τις αβεβαιότητες, για τον κοινωνικό διάλογο, ακόμα και για πράγματα τα οποία μπορεί να αμφισβητούν τις επιστημονικές μας γνωμοδοτήσεις. Είναι πράγματα όμως που είναι και αυτά σημαντικά για να είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε και με αυτούς που δεν εμπιστεύονται πάντα τις επιστημονικές μας γνωμοδοτήσεις. Να ξέρουμε γιατί, να φροντίσουμε να τις κάνουμε καλύτερες, να μειώσουμε τις αβεβαιότητες να αντιμετωπίσουμε το επιστημονικό ζήτημα που βάζει κάθε τόσο η κοινωνία μας. Και αυτό θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε την ε, στήριξή σας, τη στήριξη αυτής της Επιτροπής που είχαμε μέχρι τώρα, ότι θα συνεχίσουμε να την έχουμε και τα επόμενα πέντε χρόνια. Και φτάσαμε στο τέλος της ακρόασης. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις ερωτήσεις τους. Ευχαριστούμε την κυρία Ζασλάν Λανέλ για τις απαντήσεις της. Οι συντονιστές συνεδριάζουν στις 3 για να συντάξουν την επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αξιολόγηση της ακρόασης που μόλις κάναμε. Και στις 4 συνεχίζουμε με την Ολομέλεια της Επιτροπής μας ε, και θα έχουμε την κυρία Ζακλίν Μακλέη, την εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Θα συζητήσουμε την έκθεση για την κατάσταση και θεώρηση του περιβάλλοντος της Ευρώπης για το 2010.